Καθίστε όλοι παρακαλώ. Καταρχήν σας ευχαριστώ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Όλα ε, αυτά τα δίκτυα και οι διάδρομοι αποτελούν ε, βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών και δεδομένων των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε για να ετοιμάσουμε το σύστημα κινητικότητας του μέλλοντος, για να έχει κάποια αηφορία και βιωσιμότητα, θα πρέπει να εξετάσουμε εξονυχιστικά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στους διάφορους διαδρόμους. Γι' αυτό λοιπόν και αποτινόμαστε σε εσά ε, σήμερα, αγαπητοί Ευρωπαίοι συντονιστές, για να μας ε, παρουσιάσετε μια γενική εικόνα των σχεδίων, του συντονισμού τους, των συνεισφορών σε τι φάση βρισκόσαστε. όντω θα πραγματοποιήσουμε τη μετάβαση προς ε, σύγχρονες, βιώσιμες και έξυπνε μεταφορές. Πρόκειται να υλοποιήσουμε του στόχους μας για μεταφορές χωρίς αποκλεισμούς που θα σέβονται το περιβάλλον, θα αντιμετωπίζουν τις κλιματικές αλλαγές και θα εξασφαλίζουν καλές διασυνδέσεις. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν πρώτα να μας παρουσιάσετε το έργο σας. 7 λεπτά έχει ο κάθε Ευρωπαίος Συντονιστής και αφού ακούσουμε όλους τους καλεσμένους θα γίνει συζήτηση με τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μεταφορών. Θα ξεκινήσω πρώτα με την κυρία Άννη Γένσεν που είναι η συντονίστρια του διαδρόμου Βαλτικής Αδριατικής. Έχετε το λόγο για 7 λεπτά κυρία Γένσεν. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής Μεταφορών, αγαπητοί πρώην και νέοι συνάδελφοι, χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ σήμερα και έχω την ευκαιρία να σας παρουσιάσω το ρόλο μου και να σας παρουσιάσω και τα προσωπικά μου βιώματα και εμπειρία από, αυτό, από αυτή την θέση. Είναι, φαντάζομαι, η δεύτερη συνεδρία στην Επιτροπή Μεταφορών με τους Ευρωπαίους Συντονιστές αλλά θα ήθελα να πάρουμε μια απόσταση, να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να δούμε το ρόλο των Ευρωπαίων Συντονιστών στο όλο θέμα των διαδρόμων ε, του βασικού δικτύου. Ποια, ποιοι είναι αυτοί οι βασικοί διάδρομοι και γιατί χρειάζονται στο δίκτυο. Πρώτα αυτά τα ερωτήματα θα, θα προσπαθήσω να απαντήσω. Καταρχήν θα πρέπει να συνδέσουμε αυτή την προσέγγιση των διαδρόμων με την πολιτική των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και το μηχανισμό συνδέοντα την Ευρώπη. Πρώτα θα συνδέσω αυτά τα τρία σκέλη και μετά θα σα παρουσιάσω τον διάδρομο Βαλτικής Αδριατικής. Όπως ξέρετε, τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, τα TNT, προσδιορίζουν τα, μέτρα, τα δίκτυα μεταφορών στην Ευρώπη και η νομοθεσία αποφασίζεται, συναποφασίζεται από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συνδέονται με το μηχανισμό ΣΕΦ, σύνδετο στην Ευρώπη, που είναι ο βασικός πόρος χρηματοδότησης. Έχουμε αφενός λοιπόν την πολιτική και αφετέρου το χρηματοδοτικό μέσο, τον μηχανισμό συνδέοντα στην Ευρώπη. Και βλέπουμε πώς ε, συνδυάζονται και πώς ε, λειτουργούν αποτελεσματικά, ώστε να έχουμε έγκαιρα και αποδοτικά προγράμματα διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών με κονδύλια που θα πιάνουν τόπο. Οπότε έχουμε την πολιτική των διευρωπαϊκών δικτύων και τη χρηματοδότηση από το Συνδέοντα στην Ευρώπη. Ε, και ο συντονισμός συνδυάζει αυτά τα δύο εργαλεία. Βλέπετε λοιπόν το δικό μου διάδρομο Βαλτικής Αδριατικής και έχει διασυνδέσεις των και δύσης ε, με όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοχής και μη. Και αυτοί οι βασικοί διάδρομοι ε, καλύπτουν όλα τα μέσα μεταφορά, ε, είναι πολυτροπικοί και καλύπτουν και τι διασυνδέσει μεταξύ των τρόπων μεταφορά. Το σημαντικό όμω είναι ότι έχουν προσδώσει μια διασυνοριακή προοπτική και μια γενική πανευρωπαϊκή πολιτική στις μεταφορές. Τα... Η προσέγγιση αυτή των βασικών δικτύων ε, και των διαδρόμων έχει μια εθνική προσέγγιση των τροπολογιών και έχουμε ένα δίκτυο που φυσικά έχει διασυνοριακό χαρακτήρα, δεν σταματάει στα σύνορα. Εξού και οι επενδύσει θα πρέπει να επικεντρωθούν σε διασυνοριακά προγράμματα και θέλουμε τη δράση των συντονιστών ακριβώς για να προωθήσουμε για την έγκαιρη εφαρμογή αυτών των σχεδίων. Ε, και οι εννιά του βασικού δικτύου έχουν ένα Ευρωπαίο συντονιστή και οι Ευρωπαίοι συντονιστέ είναι οι διαμεσολαβητέ μεταξύ των κρατών μελών, των ενεχομένων και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προηγουμένω, τα κράτη-μέλη και οι ενεχόμενοι ε, συζητούν στα φόρουμ των διαδρόμων δύο φορέ το χρόνο με διοργάνωση από το συντονιστή. Πάντως, οι Ευρωπαίοι συντονιστές είναι αυτοί που επιτόπου και στο πλαίσιο του αντιστοίχου διαδρόμου του βασικού δικτύου, διευκολύνουν το διάλογο και εξασφαλίζουν το συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών. Με τα διοικητικά συμβούλια των διαφόρων προγραμμάτων και σχεδίων, με τη συμμετοχή των ενεχομένων και της κοινωνίας των πολιτών. Μάλιστα, κάνουμε και αναλύσεις, ε, μελέτες ε, για την αγορά των μεταφορών και όλα αυτά ε, τα περιλαμβάνουμε σε σχέδια εργασιών για τους εννέα διαδρόμους με αποτέλεσμα να καταλήξουμε σε, κα... σε προτεραιότητες. Είμαστε στην τρίτη γενιά τέτοιων σχέδιων εργασιών και περιμένουμε το τέταρτο σχέδιο φέτος το Δεκέμβριο και μάλιστα θα λάβετε και εσείς μέρος στην εκπόνησή του. Περνάω τώρα σε μια σύντομη παρουσίαση του δικού μου διαδρόμου, Βαλτικής Αδριατρικής. Ξεκινάει από τα από τη Βόρεια Πολωνία, τα λιμάνια της Βαλτικής, στα λιμάνια της Αδιατρικής, Σλοβενίας και Ιταλίας. Περνάει από έξι κράτη-μέλη, τέσσερα από αυτά είναι κράτη της, κράτη-μέλη της συνοχής. Και μπορεί ο διάδρομος ε, να μην έχει πολλά σημαντικά ονόματα, αλλά έχει πολύ σημαντικά και μεγάλε ευέλειε προγράμματα και σχέδια. Θα σα δώσω μερικά παραδείγματα για να σα παρουσιάσω πώ συνεργαζόμαστε με του άλλου διαδρόμου. Έχουμε καταρχήν τι διασυνδέσει τη ενδοχώρα από, ε, από το πολωνικό λιμάνι του Στέτιν και έχουμε εθνικό χαρακτήρα σε αυτά τα προγράμματα, αλλά είναι πολύ σημαντικά για τη λειτουργία αυτών των λιμανιών της Βαλτικής στην Πολωνία. Και είναι χρήσιμα και για την Πολωνία αλλά και για τις περίκλειστες χώρες όπως είναι η Τσεχία και η Σλοβακία. Ένα δεύτερο παράδειγμα αφορά το ε59, βασική σιδηροδρομική αρτηρία που συνδέει το Στέτιν με, τη, με το Βρότσοφ και την Όστροβα στην Τσεχία. Έχουν εθνικό και ταυτόχρονα ευρωπαϊκό χαρακτήρα αυτές οι διασυνδέσεις γιατί έχουν εξαιρετική σημασία και μεγάλη σπουδαιότητα για τις διασυνδέσεις μεταξύ της Τσεχίας και της Βαλτικής θάλασσας. Άλλο παράδειγμα, στην Αυστρία. Εκεί έχουμε δύο μεγάλες σύραγγες που κατασκευάζονται, Σέβεριν, με βασική σιδηροδρομική γραμμή, που είναι μεγάλη εμβέλεια προγράμματα που διεξάγει αυτή τη στιγμή η Αυστρία. 9 δισεκατομμύρια ευρώ είναι περίπου οι επενδύσεις για τα δύο αυτά σχέδια, τις δύο αυτές σύραγγες, που θα φέρουν σημαντικά ωφέλη σε αυτό τον διάδρομο. Θα μειωθεί ο χρόνος ταξιδιού και η χρήση των σιδηροδρόμων θα γίνει πιο ανταγωνιστικός. Οι σιδηρόδρομοι θα γίνουν πιο ανταγωνιστικοί. Για παράδειγμα, ε, η διαδρομή Βιέννη-Βενετία θα περιοριστεί σε ένα δύο ώρο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και από εθνική και από ευρωπαϊκή άποψη. Επίσης, το λιμάνι Κόπα στη Σλοβενία και το λιμάνι αυτό θα πρέπει να βελτιωθεί, οι διασυνδέσεις του με την ενδοχώρα να βελτιωθούν σημαντικά. Και πάλι είναι εθνικό το ζήτημα, αλλά ταυτόχρονα έχει και μια ευρωπαϊκή διάσταση. Για παράδειγμα, το λιμάνι Κόπερ είναι το πιο σημαντικό λιμάνι για την Βιέννη, για την Αυστρία δηλαδή. Οπότε είναι σημαντικό όλα αυτά τα προγράμματα να συνεχιστούν. Οι διασυνοριακές συνδέσεις είναι πολύ σημαντικές, αλλά και μερικά μεγάλες ευέλες εθνικά σχέδια είναι πολύ σημαντικά. Και νομίζω ότι έτσι θα καταστήσουμε πιο ανταγωνιστικές τις σιδηροδρομικές μεταφορές και θα μειώσουμε το αποτύπωμα διοξιδίου του άνθρακα από τις μεταφορές των φορτηγών. Ευχαριστώ. Ε, να χάσουμε χρόνο θα δώσω το λόγο στον Πάβελ, έτσι θα σας λέω. Είναι πολύ πιο απλό. Ε, είναι ο συντονιστής του διαδρόμου ε, Ρήνου Άλπεων. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω και πάλι ως Πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών και πολλά συγχαρητήρια. Μέσα σε 7 λεπτά θα προσπαθήσω να σας πω περισσότερα για το δικό μου διάδρομο ε, από το Ρήνο στις Άλπεις και να επιμείνω ε, στο πώς λειτουργεί ο διάδρομος αυτός από τη δική μου σκοπιά και πρόπτικη του γενικού ε, συντονιστού. Το πώς κυρίως μας ενδιαφέρει και όχι το τι. Βλέπετε στο χάρτη εδώ αυτό το διάδρομο Ρήνου Άλπεων. Είναι ο πιο όριμος εντό εισαγωγικών αλλά και ο πιο βραχής διάδρομος καλύπτει την πιο ανεπτυγμένη, από την πιο ανεπτυγμένη ε, γωνιά της Ευρώπης και πολύ πύκνο κατοικημένη και έχει και διάφορες προκλήσεις όπως είναι η συμφόρηση. Και αντί να συζητάμε τους κρίκους που λείπουν, ε, συζητούμε στενοπούς και συμφορήσεις και μποτιλιαρίσματα. Αν κοιτάξετε τα θέματα που μας απασχολούν, βεβαίως ε, θα πρέπει να αφαιρέσουμε αυτά στις συμφορήσεις στη Βασιλεία, ας πούμε, στο Μιλάνο, ε, το Μοντόσολα, Νοβάρα. Και να βελτιώσουμε και τη σύνδεση της ενδοχώρας με τα λιμάνια. Και όλοι έχουμε πρόγραμμα εργασίας ε, που ε, καταρτίζουν όλοι οι διαδρομοί και το εγκρίνουν τα κράτη-μέλη. Επίσης θέλουμε να προχωρήσουμε και στις συνδυασμένες μεταφορές, γιατί έχουμε το Ρήνο Έχουμε ε, τρία μέσα μεταφοράς, ε, καινοτόμες λύσεις, ε, ITS, ε, εναλλακτικά καύσιμα, το υγροποιημένο φυσικό αέριο και όχι μόνο. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για μας. Θέλουμε φυσικά να μειώσουμε το εξωτερικό κόστος ε, το σημαντικότερο είναι ο θόρυβος και οι κραδασμοί. Έχουμε ειδικέ ε, μελέτες για το πώς μπορεί να γίνει. Πολύ συχνά γίνεται συζήτηση για το θόρυβο που εμποδίζει την ανάπτυξη, γιατί οι πολίτες, ιδιαίτερα στη Γερμανία, Ε, υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες πολιτών, γελάτε όσοι είστε από τη Γερμανία, οι οποίοι έχουν πολύ έτσι, έντονες αντιδράσεις. Και φυσικά ε, αυτό που θέλουμε είναι να διατηρήσουμε την ε, κείμενη υποδομή σε καλή κατάσταση και αυτό έχει να κάνει με τις εσωτερικές πλωτές οδούς κυρίως. Εμείς ως συντονιστές προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε ε, τα χρηματοδοτικά μέσα, ε, πως είναι μια αντίστοιχη πρωτοβουλία για ε, τον αυτοκινητόδρομο ε11 στο Βέλγιο. Για να μπουν και αστικοί κόμβοι, γιατί καμιά φορά η κόμβη για τους πολίτες έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και τα, τα αρνητικά είναι ο θόρυβος, όπως είπαμε, και αυτό πρέπει να έχουμε πλατφόρμες συζήτησης για το πώς θα εφαρμόζεται ο διάδρομος και θα λειτουργεί ε, με την γενική αποδοχή του κοινού, ιδιαίτερα στους κόμβους. Αν δούμε για το πώς λειτουργούμε τώρα, αυτό είναι η επόμενη διαφάνεια, θέλω να τονίσω ιδιαίτερα στο εξής. Πώς να το πω τώρα. Ε, ε, δεν μας ενδιαφέρει μόνο το τι, το περιεχόμενο, οι κρίσιμες υποδομές, τα κρίσιμα έργα που συμφωνούμε με τα κράτη-μέλη και τις ε, τοπικές αρχές και όλους τους κατασκευαστές των project, των έργων. Αλλά το θέμα είναι πώς συνεργαζόμαστε και αυτό έχει να κάνει φυσικά με την επικουρικότητα και το δεχόμαστε, αλλά σε μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση που λαμβάνονται αποφάσεις σε διάφορα επίπεδα σε όλα τα κράτη-μέλη, άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι περίπλοκο. Και συχνά ε, είναι πολύ κατακαιρματισμένα αυτά, ε, αυτές οι αποφάσεις. Προσπαθούμε λοιπόν να φέρουμε κοντά όλους τους ενεχομένους, από πάνω προς τα κάτω, από κάτω προς τα πάνω, διαγωνίως και καθέτος να συναντώνται. Το λέει και αυτό το πρόγραμμα εργασίας, αλλά και αυτή τη στιγμή συμφωνήσουμε για κάποιες προδιαγραφές, θέλουμε και από κοινού να καλωσορίσουμε. Ας πούμε στο Ρήνο, συστήματα ενημέρωσης ε, για τα ποταμόπλια και τις μαούνες, για να σπάσει αυτή η λογική σε στεγανά ο καθένα σκέφτεται ένα κομμάτι, όχι μόνο για την υποδομή, για την ενέργεια κτλ. Ε, το βασικό μέσο είναι η πρωτοβουλία συνδέοντας την Ευρώπη, ε, διευκόλυνση καλύτερα, Connecting Europe Facility. Και είναι ένα ποσό που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για το έργο με πολύ στοχευμένες δράσεις και θέλουμε πάντα να τηρούμε τις ε, υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι ενεχόμενοι και να πιέζουμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που κάνει ανάλυση κόστους κόστους-οφέλους για όλα τα έργα. Και φυσικά εμείς αναζητούμε την ευρωπαϊκή υπεραξία ή προστιθέμενη αξία ε, και τον κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο. Αυτό είναι βασικό στοιχείο για την πρόταση για το νέο προϋπολογισμό και το σχεδιασμό των οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα θέματα που είναι διασυνοριακά χρειάζονται ιδιαίτερη έμφαση. Υπάρχει μια έννοια που σημαίνει ε, το πρόστιμο, η μορία για το, τον πρώτο κινούμενο στην πρώτη χώρα. Υπάρχουν κάποιες διασυνοριακές συμφωνίες που δεν τηρούνται. Ας πούμε όταν φτιάχνεις ένα σιδηρόδρομο και περιμένεις ε, να κάνει ε, τον υπόλοιπο κάποιος άλλος ε, σε μια άλλη χώρα και δεν ε, ολοκληρώνεται η σιδηροδρομική υποδομή. Αυτός που κάνει την πρώτη κίνηση δεν επιβραβεύεται, αλλά ε, τιμωρείται κιόλα που άρχισε να αναπτύσσει την υποδομή. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε αυτά τα θέματα σε πολύ μεγάλες λεπτομέρειε, έτσι ώστε να τηρούμε τις υποσχέσεις μας. Και για να γίνει αυτό φυσικά χρειάζεται να υπάρξει μια συμφωνία, όπως είναι το EGTC, ένας διάδρομος, μια στρατηγική. Είναι ο κεντρικός Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας. Ε, επίσης θέλουμε μια μόνο απευθυντική θηρίδα ε, για ε, το σιδηρόδρομο. Και το CCNR που είναι το Κέντρο Επιτροπής Ναυσιπλοείας στο Ρήνο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξέρει ότι ε, ε, έχει συμπληρωθεί 200 ε, χρόνια από τη λειτουργία. Να, εδώ είναι το Γκοτάρντο. Το, διάσελο είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα, όχι ευρωπαϊκό αλλά ελβετικό. Είναι η πρώτη συνδρομική σύραγγα στον κόσμο και το, το Σαν θα ανοίξει μάλλον στις αρχές του επόμενου έτους. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Προσέχετε να μην καταναλώνετε υπερβολικά πολύ αλκοόλ. Τουλάχιστον όχι εδώ σε αυτό το κοινοβούλιο. Συνεχίζουμε με την κυρία Ραντιτσόβα για τη διαδρομή της Μεσογείου. Έχετε το λόγο για 7 λεπτά. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας συγχαρώ όλους που εκλεγήκατε ή επανεκλεγήκατε ευρωβουλευτές. Ελπίζω να απολαύσετε τη ζωή σας στις Βρυξέλλες και να θεωρήσετε ότι η παραμονή σας εδώ υπήρξε επιτυχής και ότι έφερε αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια λοιπόν. Η δική μου διαδρομή, αν δει κανείς το χάρτη, η πράσινη γραμμή πηγαίνει από την Νότια Ισπανία μέσω της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Σλοβενίας, της Κροατίας, της Ουγγαρίας και μέχρι τα σύνορα της Ουκρανίας. Περιλαμβάνει πολύ σημαντικά λιμάνια, πολύ σημαντικές ε, συνδέσεις ε, οριζόντια δομών διαδρομών και αποτελεί την κύρια γραμμή από το νότο προς κάποιο άλλο μέρος της Ευρώπης. Για ποιο λόγο χρειαζόμαστε τη διαδρομή, θέλω να το επαναλάβω. Πολιτικοί λόγοι. Δεν μπορεί κανείς να μιλάει για ένωση μη συνδεδεμένη. Αν εξακολουθούμε να έχουμε ε, εμπόδια και προβλήματα στα σύνορα και πρέπει να αλλάζουμε ε, ατμομηχανές ε, στα σύνορα γιατί αλλάζει το πλάτος του σιδεροτροχιάς εγώ ως επιβάτης ε, πρέπει να περνάω από τη μια χώρα στην άλλη και το ίδιο πρέπει να κάνω και τα εμπορεύματα χωρίς να υπάρχει κανένας φραγμός. Ομαλά, γρήγορα και αποτελεσματικά. Πολιτική λοιπόν η λόγια. Για να έχουμε μια ένωση σημαίνει μια ένωση ε, συνεπάγεται ότι είμαστε συνδεδεμένοι και υλικά. Επίσης, οικονομικοί λόγοι. Κάθε άρση φραγμού σημαίνει περισσότερο εμπόριο, περισσότερες μεταφορές. Για να έχουμε όλο και περισσότερες μεταφορές, δεν μπορούμε να τους βάζουμε συνέχεια τρικλοποδιές. Δεν μπορούμε να τα μεταφέρουμε συνέχεια όλα με φορτηγά. Έχουμε παραμείνει στα ίδια και στα ίδια. Δεν κινείται τίποτα. Υπάρχει κατάρρευση απόλυτη. Ε, στους αυτοκινητοδρόμους μας η συμφόρηση είναι τρομακτική διότι οι μεταφορές αυξάνονται σε τέτοιο βαθμό μέσω φορτηγών, μέσω αυτοκινητοδρόμων και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό στην καθημερινότητα. Όλοι συμφωνούμε ότι αυτό περιπλέκει τις ζωές μας. Δεν βοηθά να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής μας. Τελευταία φορά εγώ που έζησα να περνάω τη Γαλλία 5.000 ε, χιλιόμετρα, η Γερμανία, ξέρετε, προσπάθησε να λύσει αυτό χτίζοντας έναν τρίτο αυτοκινητόδρομο για να ε, ε, πρόσθεσε μάλλον μια λωρίδα στους αυτοκινητοδρόμους για να έχει όλο και περισσότερα φορτηγά. Το θέμα είναι ότι σε 30 χρόνια έχουν μπει όλο και περισσότεροι περισσότερα φόρτηγα. Χρειαζόμαστε περισσότερε μεταφορέ στου σιδηροδρόμου, οι οποίοι είναι περιβαλλοντικά πιο φιλικοί. Θέλουμε πραγματικά να συνδέσουμε δηλαδή την Ευρώπη με περιβαλλοντικά φιλικές συνδέσεις. Σε αυτόν το διάδρομο λοιπόν θα ήθελα να σας δείξω κάτι που θα πρέπει να προσέξετε, τα εμπόδια, τα προβλήματα και σας παρακαλώ να υποστηρίξετε και να βοηθήσετε. Ποιε είναι λοιπόν οι δυσκολίε τι χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε. Θα ήθελα να τονίσω ότι αυτή, η διαδρομή έχει τα περισσότερα έργα. 142 το αριθμό. Συνολικά 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι πραγματικά μεγάλο έργο στο σύνολό του. Αναθρήσει κανείς όλα τα επιμέρους έργα. Αυτό όμως που χρειαζόμαστε πραγματικά είναι το εξή. Πρώτον, βελτιώσεις ε, στη διέρευση των συνόρων μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας, ειδικότερα στη σύνδεση Βαρκελόνης-Μομπελιέ. Αύριο θα συνεδριάσει μια ομάδα εργασίας που δημιουργήσαμε με τους εταίρους από αμφότερες τις πλευρές, ε, από τη Γαλλική και την Ισπανική, για να γίνει κάποια διαπραγμάτευση με μια προσπάθεια, σε μια προσπάθεια να λυθούν κάποια προβλήματα, να αρθούν τα εμπόδια ούτως ώστε να ολοκληρωθούν οι συνδέσεις σε αυτή την περιοχή. Όλοι το επιθυμούν. Πέρυσι συναντηθήκαμε για πρώτη φορά. Αλλά χρειάζονται και άλλα βήματα για να ολοκληρωθεί. Ζητά συγγνώμη, μιλήτρια second, please. Sorry. I think that we are very successful in connection trees, Ljubljana, Zagreb, Budapest. Ljubljana Zagreb και Βουδαπέστη έχουμε ήδη μια επιτυχή σύνδεση και έχουμε σημειώσει βαθιά πρόοδο σε σχέση με τη σύνδεση Κόπερ Βάτσα. Το βασικό τα μεγαλύτερα ερωτηματικά υπάρχουν στη σύνδεση Λιών Τωρίνου. Ατέρμονη συζήτηση. Για μένα, 30 χρόνια πια γίνεται αυτή η συζήτηση. Από το 1990. 400 εκατομμύρια ευρώ έχουν δαπανηθεί για την ανάλυση κόστους και ωφελών του έργου αυτού, τη σύνθεση αυτής Λιών Τωρίνου. Χιλιάδες σελίδες έχουν γραφτεί με ελέγχους, αξιολογήσεις, εκτιμήσεις. 20 χρόνια συζητούσαν αν πρέπει να γίνει ή όχι. Και όταν τελικά κατάληξαν σε μια συμφωνία, είπαν είναι σαφέ σε σχέση κοστοφέλους, είναι λίγο ψηλότερο λόγω περιβαλλοντικών αιτιών, παρόλα αυτά θα το κάνουμε. Σήμερα, όταν λέω εμείς, ενώ η, εθνική, η κυβέρνηση της Ιταλίας, η κυβέρνηση της Γαλλίας, και άλλες 25 κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή υπάρχει ευρεία συνένεση, ευρεία συμφωνία. Εγώ έχω πάει εκεί πολλές φορές γιατί είναι κάτι που με αφορά και είναι διαφορετικό να πηγαίνει κανείς να το βλέπει από ότι να διαβάζει σελίδε. Χθε είχαμε την για την, τα εγκαίνια για τα πρώτα 9 χιλιόμετρα του διαδρόμου. Σκοπός είναι να μειωθεί ο αριθμός φορτηγών στους αυτοκινητοδρόμους σημαντικά. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω αριθμούς, να, να σας εξηγήσω για πόσους τόνους διοξιδίου του άνθρακα μιλάμε, τι απαλλαγή από ανθρακούχε εκπομπέ. αλλά εμείς είμαστε εδώ που είμαστε, έχουν συμφωνήσει οι κυβερνήσεις, τα κοινοβούλια Γαλλία και Ιταλία. έχουν ξανά συμφωνήσει και ξανά και ξανά και συνεχίζουμε. Αν έχετε ερωτήσεις Ευχαριστώ να τις απαντήσω, αλλά Ο δρόμο του μεταξιού θα φτιαχτεί πιο γρήγορα από ότι να φτιάξουμε εμεί μία σύραγγα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, καλεσμένο μα, ο κύριο Πατ Κόξ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ. Σας συγχαίρω όλους τα οικία πρόσωπα, αλλά και τους συναεκλεγέντες ευρωβουλευτές. η ενημέρωσή σας ε, αποτελεί σημαντικό τμήμα των καθηκόντων μου και χαίρομαι που έχω αυτή την ευκαιρία στην αρχή της θετίας. Εγώ θα σας μιλήσω για το διάδρομο Σκανδιναβίας Μεσογείου. Περνάμε στην επόμενη διαφάνεια. Βλέπετε τα διάφορα πολύχρωμα κουτιά. Κάθε κουτί είναι και ένα κράτο. Έχουμε τη Φιλανδία, τη Σουηδία, τη Δανία, τη Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία και Μάλτα. Και επίση, ε, ανώ αριστερά έχουμε την Νορβηγία που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Είμαστε ο μακρύτερο ε, διάδρομο από τους εννέα γεωγραφικούς διαδρόμους. Καλύπτουμε 9.600 χιλιόμετρα σιδηροδρόμου, 6.400 χιλιόμετρα οδικών αρτηριών. Έχουμε 91 κόμβους, πολυτροπικότητα. Έχουμε 44 λιμάνια, 45 ε, τερματικά, 29 ε, ε, τέτοιες αστικές ζώνες και έχουμε δύο βασικά σχέδια, BBT, το, η κεντρική σειρά του Μπρένερ και το FBFL που είναι ο πάγιος σύνδεσμος δύο νησιών, Φέμαν και Λόλαντ. Επίσης, έχουμε 15% πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν σε αυτό το διάδρομο πριν από το Brexit. 16, αν γίνει τελικά, 16,8% της απασχόλησης και 20% του ευρωπαϊού ΑΕΠ. Ε, και η μόνη χώρα συνοχής είναι η Μάλτα από αυτές. Τώρα, περνάμε ε, στο παγιο σύνδεσμο των ίσων Φέμαν και Λόλαν. Θα έχουμε την ε, μεγαλύτερη υποβρύχια σύραγγα που θα συνδέει τη Δανία και τη Γερμανία 18 χιλιόμετρα θα είναι το μήκος της και θα εξαλείψει ένα ε, βασικό πω σημαντικό σημείο συμφόρησης και περιμένουμε να ολοκληρωθεί μέχρι το 2028. Το κόστος κυμαίνεται γύρω στο 7,1 δισεκατομμύρια ευρώ. 40% θα προέλθει από ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση, όχι για τα πάντα, μόνο για το σιδηροδρομικό σκέλος, ενώ το οδικό σκέλος ε, θα, θα χρηματοδοτηθεί από διόδια και χρηματοδότηση χρηστών. Και θα μειώσει αισθητά την διάρκεια του ταξιδιού και την απόσταση κατά 160 χιλιόμετρα θα μειωθεί η απόσταση, ο χρόνος θα μειωθεί κατά μια μισή ώρα. Επίσης, εμ, θα συνδέσει τη Κοπεχάγη με το, με το Αβούργο, το Γκέτεμπορκ, το Όσλο με τη Στοκχόλμη. Σημαντική, σημαντικό το σχέδιο αυτό και συνήθω όταν έχουμε ένα σχέδιο μεταφορών έχουμε μια βραχυπρόθεσμη προοπτική. Όταν όμως ε, έχουμε τέτοιους συνδέσμους όπως ε, υποβρύχες ε, σύραγγες για τα νησιά Θέμα και Λόλαντ έχουμε πραγματικά μια πολύ ευρύτερη προοπτική και φυσικά θα συμβάλλει στην απαλλαγή μα από τι εκπομπέ άνθρακα. Και πάμε σε ένα άλλο σημαντικό ε, σχέδιο μεταξύ Αυστρίας και Ιταλίας, τη σειρά Γκαμπρένερο. Ε, είναι, θα, ε, είναι ένα χιλιόμετρο περίπου κάτω από την κορυφή του βουνού Μπρένερο και θα είναι το μακρύτερο, η μακρύτερη σύραγγα του κόσμου. θα πάρει το ρεκόρ από τον Κόταρτο και ένα σημαντικό τμήμα μέχρι το 2028 θα έχει ολοκληρωθεί. Μέχρι στιγμής έχουμε ε, ολοκληρώσει την εξκαφή 109 από τα 230 χιλιόμετρα. Ε, μάλιστα, 3, θα τέταρτα θα είναι διαρευνητικές σύραγγες για να αντιληφθούμε την υδρολογία και την ε, κατάσταση γεωφυσική και το 1 τέταρτο είναι βασικό. Ε, 1 τέταρτο είναι το ε, κεντρικό τούνελ που έχει ολοκληρωθεί και περιμένουμε μέχρι τα τέλη του 2028 να ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις και να έχουμε, ήδη θα έχουμε πολλές ε, μηχανές ε, που λειτουργούν με 40% ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Το κόστος γύρω στα 8,7 δισεκατομμύρια, 40% ξεχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση που ίσως ανέλθει στο δεύτερο, δεύτερη φάση του μηχανισμού συνδέοντας στην Ευρώπη. Πάντως Μέχρι στιγμής έχουμε δώσει 2 δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Συγχρηματοδότηση, το, το υπόλοιπο 30% από την, θα προέλθει από την Ιταλία και 30% από την Αυστρία. Επίσης έχουμε σημαντική αύξηση της δυναμικότητας ε, και φυσικά πολυτροπικότητα. Έχουμε σημαντικό πρόβλημα με τη διεύρυ... με το διέλευση του Μπρένερο. 2,4 εκατομμύρια φορτηγά. Πολύ αρνητικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο και δεν υπάρχουν εναλλακτικέ λύσει αυτή τη στιγμή. Αυτή η σύραγα του Μπρένερο θα είναι η εναλλακτική λύση. Επίση, ένα τόνο εμπορευμάτων με θερμοδρομικέ μεταφορέ έχει πολύ, λιγότερο, ε, πολύ λιγότερε εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα από τον αντίστοιχο τόνο στι οδικέ μεταφορέ. Οπότε είναι πολύ σημαντικό. Και θα ήθελα να κάνω και μερικά γενικά σχόλια. Στο δικό μας διάδρομο έχουμε καινοτομήσει ώστε να περάσουν οι συστάσεις των εμπειρογνωμόνων σε ένα εργαστήριο ιδεών, ώστε πραγματικά να έχουμε έξυπνες μεταφορές. Αυτό είναι σημαντικό τμήμα και σίγουρα οι Βρυξέλλες δεν ξέρουν τα πάντα, αλλά έχουμε πολύ σημαντικούς εμπειρογνώμονες και επιτόπου, που όμως μερικές φορές είναι απομονωμένοι προωθούμε τις βέλτιστες πρακτικές μεταξύ ομοτήμων, χρησιμοποιούμε συστάσεις και επίσης ε, έχουμε ε, εξετάζουμε και την οικονομική ε, συνεργασία των λιμένων. Το κάναμε και για τα αεροδρόμια και για τους αστικούς κόμβους, ώστε να έχουμε το car sharing, τα ηλεκτρικά οχήματα, την μείωση τον εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα με τη χρήση ποδηλάτων, τη συμβολή και του περπατήματο. Επίση, ε, σιδηροδρομικέ μεταφορέ και ανάλυση του έχει γίνει τρει φορέ. Πολύ περίπλοκο, ε, πολυσύθετο θέμα, αλλά πραγματικά με το διάδρομο αυτό θα συμβάλλουμε τα μάλα. Επίση, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείριση τη Κυκλοφορία, το ERTMS, ε, τη Σιδηροδρομική κυκλοφορία, θα βελτιώσει τη, τη δυναμικότητα των νέων συστημάτων. Έχουμε λοιπόν ένα εργαστήριο ιδεών και για τις ιδεονομικές μεταφορές επιβατών και θέλουμε να προωθήσουμε τις φιλοπεριβαλλοντικές δημόσιες συμβάσεις. Είναι σημαντικό θέμα της δημόσιας πολιτικής. Επίσης, για τις ανακοινώσεις. Έχουμε πολλές κυβερνητικέ δομές, δεν θα επισέλθω σε όλες αυτές. Ε, θεωρούμε ότι είναι χρήσιμες έγκαιρες ε, σε πρώιμη φάση ε, διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερομένους. Έχουμε τακτικές συναντήσεις με βασικούς ε, συμμετέχοντες ε, συναντήθηκα με ε, δημάρχους των περιοχών γύρω από τον Μπρένερο και θέλω να έχω τακτικές επαφές μαζί τους, τον έχω ιδιαίτερο συμβασμό και μάλιστα τα τελευταία χρόνια είχαμε 100.000 επισκέπτες, τεράστια υποστήριξη, θετική, ανοιχτής πόρτες, ανοιχτό μυαλό, ανοιχτή επικοινωνία είναι τα βασικά μας χαρακτηριστικά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κόξ για όλα αυτά που μας είπατε για τον περιβόητο διάδρομο της Μεσογείου. Ε, θα ανοίξω τη συζήτηση. Δεν κρατιέστε, κάνετε τις ερωτήσεις. Η κυρία Τάλερ είναι πρώτη. Έχετε το λόγο. Παραλέγω να πω, έχετε το αυτοκίνητο. Εν πάση Ευχαριστώ. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Πατ Κόξ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση κύριε Κόξ και χαίρομαι πάρα πολύ που μας λέτε για προόδους και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το πάθος με το οποίο μιλήσατε για το, ε, τη σύρεγγα αυτή ε, της βάσης του Μπρένερου. Δεν έχουμε εναλλακτική λύση, το είπατε κι εσείς. Και εγώ από εκείνη τη γωνιά της Ευρώπης προέρχομαι και μας τελειώνει και ο χρόνος. Τουλάχιστον έχω την αίσθηση ότι δεν έχουμε χρόνο. Έχουμε 2,5 εκατομμύρια ε, φορτηγά που πηγαίνουν από τη Γερμανία στην Ιταλία από τον Μπρένερ και ε, περιμένει ο πληθυσμός εκεί αυτή η επένδυση δισεκατομμυρίων να οδηγήσει και σε μια αισθητή μεταφορά της κυκλοφορίας από τον αυτοκινητόδρομο στο σιδηρόδρομο. Υπάρχει κατάλογος. Ε, υπάρχει κατάλογος. Γι' αυτό... Έχετε ένα πρόγραμμα δράσης με συγκεκριμένα ορόσημα για να μπορούμε να συζητήσουμε και πόσο κοστίζουν αυτά τα γραφειοκρατικά εμπόδια για τις καθυστερήσεις και τα διάφορα τεχνικά προαπαιτούμενα. Γιατί θα εξαρτηθεί πάρα πολύ ε, και από τη σοβαρότητα, την ταχύτητα με την οποία προχωρούν τα γειτονικά κράτη. Παρακαλώ να μην παρεξηγηθώ. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε κανέναν, αλλά μιλούμε για χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων, μεταξύ άλλων. Και αν δεν υπάρχει ταυτόχρονος ε, συντονισμός, τότε μας κοστίζει αυτό και χρήματα των φορολογουμένων, αλλά και αξιοπιστία. Έχετε διδάγματα για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ. Προσπαθήστε να σέβεστε το χρόνο σας, 1,5 λεπτό έχετε έκαστος, γιατί πιέζουν πάρα πολύ χρόνοι. Ο κύριος Ντάνιελσον, για ένα λεπτό. Thank you. Ε, Ευχαριστώ όλους σας για τις παρουσιάσεις σας. Έχω μια γενική ερώτηση, αφορά όλους σας. Αν μπορούσατε να δώσετε μία γενική συμβουλή όχι να αφορά το δικό σας ε, έργο μόνο, στον επόμενο ή την επόμενη επίτροπο, ούτω ώστε να επιτύχουμε τους στόχους TNT, αλλά και να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μέχρι το 2030. Ποια συμβουλή θα ήταν αυτή και μετά για τον κύριο Κόξ. Έχω μια ερώτηση για τον διαδρομό ε, Σκανδιναβίας-Μεσογείου. Σε όλα αυτά τα δίκτυα φυσικά υπάρχουν περιφερειακές συνεργασίες που έχουν ξεκινήσει, ούτω ώστε να ολοκληρωθούν τα δικά τους τα επιμέρους τμήματα των δικτύων. Ε, το παράδειγμα που έχω στο νου μου είναι το δίκτυο τοπικών και περιφερειακών ε, αρχών μεταξύ Αμβούργου και Όσλο για το βόρειο τμήμα του διαδρόμου. Και όταν λέω εκπρόσωποι αυτής της συνεργασίας, εννοώ ότι εξακολουθούν να έχουν προβλήματα όσον αφορά τη σχέση τους με την κυβέρνηση και με το διάλογο με την κυβέρνηση και ότι οι υποδομές σταματούν στα εθνικά σύνορα και η ερώτησή μου είναι, συμφωνείτε με αυτή την εικόνα και σε τι θα δίνατε προτεραιότητα αν ήταν να βάλουμε πίεση στις κυβερνήσεις ούτως ώστε να επιληθεί αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε. Κύριε Μπαουσά, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ καταρχάς ε, τους ομιλητές και τους τέσσερις για τις ε, παρεμβάσεις τους. Πολύ πρακτικές. Ε, θέλω να αναφερθώ σε κάτι συλλογικά. Δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι οι διάδρομοι είναι οι υποδομές που δείχνουν στους πολίτες πόσο σημαντική είναι η Ένωση και η Ευρώπη και ευκαιρίες που μας δίνει η Ευρώπη γιατί δεν έχουμε 27 κατακαιρματισμένους χώρους, αλλά ένα ενιαίο χώρο, κοινό. Πολλές φορές ακούμε ότι από τους διαδρόμους εποφελούνται μόνο οι περιφέρειες, ε, οι άμεσα ενδιαφερόμενες. Στην Ισπανία, ας πούμε, μόνο η Βαλένθια για να στέλνει τα πορτοκάλια ε, παντού στην Ευρώπη από τον Μεσογειακό διάδρομο. Ή η Καντάβρια για να στέλνει το γάβρο και τις αντσούγες ε, σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν όμως και ε, άλλες απομακρυσμένες περιφέρειες που είναι στο κέντρο της χώρας, όπως είναι η Ριόχα, ας πούμε, που είναι ανάμεσα σε δύο διαδρόμους, το Βόρειο και το Μεσογειακό, και μπορεί να στείλει τα κρασιά της και στο καλύτερο εστιατόριο στην Ευρώπη, όπως και τα άλλα προϊόντα της Ευρώπης να έρχονται σε εμά. Τι εννοώ, γιατί τα λέω όλα αυτά ε, για τις απομακρυσμένες περιφερειακές περιφέρειες. Αν έχουν καλύτερες υποδομές, θα βελτιωθούν οι εισαγωγές, εξαγωγές, η απόδοση και όχι μόνο. Οι ε, πολίτες θα αισθάνονται περισσότερο Ευρωπαίοι από ποτέ και είναι κοινή ευθύνη μας αυτή. Ε, συγχαρητήρια για τις παρουσιάσεις και θα πρέπει όλοι να έχουμε επίγνωση του σπουδαίου έργου ε, που σημαίνουν όλοι αυτοί οι διάδρομοι για την Ευρώπη. Ευχαριστώ από τους πράσινου, η κυρία Ντεπαχνέ. Ναι. Ευχαριστώ για την εστίαση που δίνεται στη δεσυνοριακή διάσταση ε, ε, είναι πολύ σαφές αυτό και κοινή μας ε, εστίαση και ιδιαίτερα η απομάκρυση από το διοξίδιο του άνθρακα. Έχω μια ειδική ερώτηση. Κυρία Γένσε, είδαμε πολλά μικρά αεροπλάνα στην παρουσίασή σας στο χάρτη και ως πράσινη κάπως στραβοκατάπια. Ποιο είναι το ποσοστό που δίνεται σε κάθε μέσο μεταφοράς, ενώ το χρόνο και τα χρήματα που αφιερώνεται, γιατί στις συνδυασμένες μεταφορές θα πρέπει να είναι συνδυασμένες, να κοιτάμε περισσότερο το σιδηρόδρομο, ακόμα και αν είναι δύσκολη η υποδομή, γιατί θέλει και υπομονή για να φτιαχτεί όλο το δίκτυο, ενώ πιο εύκολο εκ πρώτης όψεως είναι να χτίσεις ένα αεροδρόμιο. Αλλά οι στοδυνικές δεν είναι το καλύτερο για το κλίμα, χρειάζεται καλές συνδυασμένες μεταφορές και θέλω να μου το απαντήσετε. Κύριε Βοητσεχόφσκι, και ελπίζω να μην το πολύ σκότωσα, ε, για τις εσωτερικές πλωτές οδούς και με την κλιματική αλλαγή ταυτόχρονα υπάρχει ανάγκη να ασχοληθούμε περισσότερο και να αναπτυχθούμε περισσότερο προς τις πιο ουδέτερες ως προς το διοξίδιο του άνθρακα δυνατότητες. Έχουμε όμως και τη λειψιδρία και αυτό μειώνει τη στάθμη των ποταμών. Αυτό επηρεάζει τη δουλειά σας. Χρειάζεται προσαρμογές. Το έχετε σκεφτεί. Και έχω και μια ε, πολύ τοπική ερώτηση για τη δική μου εκλογική περιφέρεια. Με το, τη Στουτγάρδη Ούλμ ε, ε, υπάρχει υπερταχεία και στις μεταφορές επιβατών. Αλλά τι γίνεται με τις εμπορευματικές μεταφορές. Και προς τον κύριο Κόξο θέλω να ρωτήσω για τις συνδυασμένες μεταφορές γιατί ανάλογα με τους διάφορους ενεχόμενους αναχώρα αυτοί ανήκουν σε διαφορετικούς φορείς ε, ε, για την απαγκίστρωση από το διοξίδιο του άνθρακα. Πώς ε, μπορείτε εκεί να συγκεράσετε τις απόψεις. Και για το Λιόν το Ρήνο θέλω να ρωτήσω την Αλκυρία πόσο ποσοστό από τον προπολογισμό σας πήγε σε αυτό το έργο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Προσπαθείτε παρακαλώ να ε, σέβεστε το χρόνο ε, ώστε να μπορούν να μιλήσουν και οι συνάδελφοι. Κυρία Λεσόντα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Προς την κυρία Ρεντικόβα ήθελα να πω ο διάδρομος της Μεσογείου είναι ο βασικός άξονας Ανατολής Δύσης στα διευρωπαϊκά δίκτυα κάτω από τις Άλπεις. Θα πρέπει να αποτελεί μια σύνδεση συνδυασμένων μεταφορών από τη Δυτική Μεσόγειο μέχρι το κέντρο της Ευρώπης. Θα πρέπει να συμμετάσχει με οδούς και συνδρομικές οδούς σε σημαντικά κομμάτια όπως η Άλπης και η Μεσόγειος. Και όπως είπατε πριν λίγο, έχουμε τόσο μεγάλη αύξηση ε, διπλασιασμό σε 30 χρόνια των οδικών μεταφορών και αυτό οδήγησε σε ε, μείωση των σιδηροδρομικών μεταφορών ε, στη Γαλλία. Στο Περπινιό Γανζής ε, έχουμε μια διαδρομή που καταργήθηκε και βλέπουμε ξαφνικά 25.000 ε, επιπλέον φορτηγά κάθε χρόνο στους γαλλικούς αυτοκινητοδρόμους. Το έργο είχε σκοπό να μειώσει τα φορτηγά στους δρόμους μας, ενώ συμβαίνει το αντίθετο σύμφωνα παρά τα εκατομμύρια που δαπανήθηκαν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Πιο γρήγορα τώρα. Ο κύριος Ρικέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λακωνικά. Θα ήθελα να χαιρετήσω καταρχήν και τους τέσσερις συντονιστές μας. Ε, παρακολουθήσατε τη νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα έξυπνα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών που στόχο έχουν να, πλουστεύσουν και να μειώσουν τις γραφειοκρατικές διατυπώσεις, τις προθεσμίες, το κόστος, τις καθυστερήσεις. Έχετε γνώση αυτής της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχετε κάποιες παρατηρήσεις από αυτού. Μία ερώτηση και προς τον Πατ Κόξ για, το, για τη σύραγγα του Μπρένερου. Τι γίνεται με την ε, γερμανική πλευρά. Οι πρόσφατες δηλώσεις ε, της Καγκελαρίου για ε, τα 100 δις τις επενδύσεις ε, στο σιδηρόδρομο δεν θα εκτρέψουν τον, τη σύραγγα και προς την γερμανική πλευρά. Επίσης, τι γνώμη έχετε για την γαλλική πρόσβαση στη σύραγγα Λιών του Ορίνου. Όχι για το ίδιο το έργο, αλλά για τα 80 χιλιόμετρα πριν από τη σύραγγα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λιμπεράτσκι. Δύο γενικές παρατηρήσεις. κάθε αύξηση 1% του ΑΕΠ ε, απαιτείται περισσότερες μεταφορές. Θα έλεγα ότι ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά όχι απολύτω. Εγώ θα έλεγα ότι κάθε βελτίωση στι μεταφορέ μα δίνει τη δυνατότητα για αύξηση και το ΑΕΠ. Και με τις μεταφο... χωρίς μεταφορές δεν πρόκειται να έχουμε ε, ενίσχυση και του ΑΕΠ. Επίσης, έχουμε τη βασική τριάδα, διευρωπαϊκά δικτύα, το μηχανισμό σύνδετος στην Ευρώπη και τους ε, ειδικού αυτούς διαδρόμους. Ευχαριστώ για αυτή την τριάδα που μα επισημάνατε και που την αναδείξατε. Και κυρία Γένσεν. Εγώ είμαι ο παλιός σας φίλος, όχι εσείς. Ε, και πιο ηλικιωμένος. Τι γίνεται με το ποταμό Όντερ, το διάδρομο του ποταμού αυτού. Έχει παραμεριστεί τελείως και έχετε σκεφτεί την πιθανότητα ρυθμίσης όχι μόνο για το ποταμό Όντερ, αλλά να έχουμε συστήματα έξυπνων μεταφορών και εφαρμογές και κατά μήκος αυτού του διαδρόμου. Και θα έλεγα ότι ο διάδρομος που συντονίζει η κυρία Γένσεν ε, είναι πολύ επιτυχημένος και μάλιστα 400 χιλιόμετρα αυτού διαδρόμου περούν από τη δική μου εκλογική περιφέρεια, οπότε γνωρίζω ε, από πρώτο χέρι πόσο αποτελεσματικοί είστε. η κυρία Γκαρσία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους για τις ομιλίες σας. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να εκφράσω την ικανοποίησή μου προς την κυρία Ρεντίκοβα για το ότι συμπεριλήφθηκε και η Σαραγώσα στο βασικό μεσογειακό διάδρομο για την περίοδο 2021-2027. Ε, όπως ξέρετε και η, Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε πόσο σημαντικό είναι να συνενώσουμε την αντιδρατική πλευρά με τη Μεσόγειο γιατί μας δίνουν διεξόδους προς την Αμερική και την Αφρική και γι' αυτό είμαι πρόθυμη να συνεργαστώ μαζί σας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με όλου του ενδιαφερόμενους ώστε να προωθήσουμε το σχέδιο αυτό για να ε, λάβει σάρκα και ωστά κάποια ημέρα παρόλο που πραγματικά φαίνεται τιτάνιο έργο. Τώρα, προς τους τέσσερις συντονιστέ μας θα ήθελα να σταθώ σε κάτι που είπε ο κύριο Σέκη, ο συνάδελφο στι αρχέ του Σεπτεμβρίου. Ο κύριος Σέκη μίλησε για την σημασία που έχει η καλύτερη και αποτελεσματική ενσωμάτωση του κεφαλαίου και χρηματοδότησης για τα διάφορα σχέδια και προγράμματα των ευρωπαϊκών δικτύων. Θα πρέπει να δούμε πώς θα κινητοποιήσουμε, πώς θα προσελκύσουμε περισσότερα κονδύλια από πολλούς ενδιαφερόμενους. Ποια είναι η δική σας γνώμη, τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε για να προσελκύσουμε περισσότερα κεφάλαια και χρηματοδότηση για τα σχέδια αυτά. Επίσης, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσει ε, τη έκθεση για τον εξορθολογισμό των μέτρων ώστε να προωθήσουμε την ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το Φεβρουάριο του 2019 μια πολύ θετική έκθεση με ξεκάθαρη ε, ευρωπαϊκή προοπτική και όραμα με συγκεκριμένα με συγκεκριμένες προτάσεις όπως Ευρωπαϊκή Αρχή για τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρία Μπιλμπάου, αντίκα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις. Πολύ σύντομα, μερικές ερωτήσεις για όλους τους συντονιστές. Ακούσαμε σε προηγούμενη ακρόαση τους συντονιστές των υπολείπων έργων. Εσείς που εργάζεστε σε αυτά, μιλήσατε για το πρόβλημα των παραμεθόριων περιοχών. Πόσα έχουμε λύσει στα προγράμματα προτεραιότητας, καμία. Εγώ κατάγομαι από τη χώρα των Βάσκων, όπου στην Ισπανία έχουμε προβλήματα με τα ε, σύνορα Ισπανίας-Γαλλίας και είναι ο άξονας της Μεσογείου αλλά και του Ατλαντικού. Αλλά αυτό επανέρχεται και στα άλλα σύνορα. Τι μπορούμε να κάνουμε για να υποχρεώσουμε τα κράτη-μέλη να σέβονται την προθεσμία το 2013 κάναμε αναθεώρηση, είναι σαφή τα ε, έργα. Το ελεγκτικό συνέδριο έβγαλε μια έκθεση που ε, εντοπίζει και ανοιχνεύει αυτό που λέγαμε εμεί, την κακή διαχείριση των πόρων από τα κράτη-μέλη και τελικά δεν έχουν εκτελέσει με συνέπεια τα προγράμματα και τα έργα, γι' αυτό δεν είμαστε συνδεδεμένοι. Και αυξάνονται τα φορτηγά και πληθύνονται οι ε, εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα στα σύνορα. Στους διαδρόμους σας θα ε, φτάσουμε ε, να καλύψουμε τις προθεσμίες και εγκαίρως σε λειτουργία ή θα έχουμε και νέα αναθεώρηση. Πιστεύετε ότι μπορούν να προσθεθούν και άλλα έργα χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί αυτά που τρέχουν από το 1994. Πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Γιατί θα πρέπει να τολμήσετε να πείτε ότι τα κράτη-μέλη δεν εκτελούν με συνέπεια τα έργα αυτά. Και γι' αυτό δεν είναι περίεργο που η Γκρέντα Τούμπερκ ηγείται σε αυτό ε, το κίνημα και καταγγέλει τους πολιτικούς ότι δεν συνεισφέρουν στη μείωση των εκπομπών. Γιατί όλοι καθημερινά βλέπουμε τη συμφόρηση την κυκλοφοριακή ε, στα σύνορα και στους διάφορους αυτοκινητοδρόμους. Βγείτε δημόσια και τολμήστε να πείτε ε, τι τρέχει, να καταγγείλετε τα κράτη-μέλη και θα με έχετε στο πλευρό σας. Ευχαριστώ. Περίπου τηρήσατε το χρόνο σας, ενάμιση. Εντάξει. Allez, monsieur Fidanza, je compte sur vous. Ο κύριο Φιντάντσα, ενάμιση λεπτό, εσείς θα το τηρήσετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα δοκιμάσω τέσσερα σημεία στα γρήγορα. Κυρία Ραντικόβα, είπατε ότι το τωρινό Λιόν δεν τελειώνει ποτέ. Συμφωνώ. Φαίνεται ότι ξαφνικά, επιτέλους μετά από απαράδεκτε καθυστερήσεις ετών, προχωράμε στο σωστή οδό. Χθε εγκαινιάστηκαν τα πρώτα 9 χιλιόμετρα, στα οποία αναφερθήκατε, αλλά για την τωρινό Λιόν και για τον Μπρένερ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον συντονιστή τι μπορεί να γίνει από την Επιτροπή μας για να σας βοηθήσουμε να επιταχύνετε τους χρόνους εργασιών. Δεύτερο θέμα, το μηχανισμός συνδέοντας την Ευρώπη έχει αποδείξει ότι λειτουργεί σωστά με καλά αποτελέσματα. Θεωρείτε ότι μπορεί να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του να συντονιστεί καλύτερα το CEF με άλλα ταμεία του InvestEU, για παράδειγμα, άλλοι πόροι που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο. Τρίτη και τέταρτη ερώτηση μαζί αναφέρατε ξεχωριστά Βοητσεκοσκή και Κόξ το θέμα των εναλλακτικών εγώ ήμουν συντονιστής, ε, ε, ε, εισηγητής της σχετικής έκθεσης και το TMS. Τι μπορούμε να κάνουμε για να αυξήσουμε τις επενδύσεις και την υλοποίηση αυτών των σημαντικών δύο πυλώνων που θα βοηθήσουν να γίνουν πιο βιώσιμοι και πιο ασφαλείς οι διάδρομοι αυτοί. Ευχαριστούμε. Κύριε Ομγκριν, έχετε το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους σας. Πολύ ενδιαφέρουσα. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσιάση. Αναφέρατε ειδικότερα την απαλλαγή από ανθρακούχε εκπομπέ, αλλά για να, για να καλύψουμε τις, ε, τους στόχους του Παρισιού πρέπει να... Συγγνώμη, δεν ακούμε σωστά τη μετάφραση, την διερμηνία. Η γαλλική καμπίνα. Εντάξει, ωραία. συγγνώμη. Να ξεκινήσω από την αρχή. Ωραία, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους σας. Πολύ ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις, ειδικότερα αναφέρατε όλη την ανάγκη απαλλαγής από ανθρακούχες εκπομπές. Για να επιτύχουμε τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού, χρειάζεται 100% απαλλαγή του συστήματος μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ανθρακούχες εκπομπές. Από δική σας εμπειρία, ποια είναι τα κύρια εμπόδια για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Ευχαριστούμε πολύ. Σαφές και σύντομο, κύριε Τι, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, μια ερώτηση προς τον Πατ Κόξ. Επειδή ε, ως φιλελεύθερο μέλος του Κοινοβουλίου από τη Βόλια Γερμανία ήθελα να μάθω θα γίνει πραγματικότητα γρήγορα. το Μπέλτο διότι είναι σημαντικό και για τη σκανδιναβική περιοχή ε, Κοπενχάγη, αυτή η περιοχή προς το Αμβούργο που έχει το τεράστιο λιμάνι, οπότε η ερώτησή μου είναι, επειδή πιστεύω ότι έχουμε το πρόβλημα στο Μπρένερ και στο Φιμεμπέλτ, ότι οι διαδικασίες της Γερμανίας δεν είναι αρκετά γρήγορες σε σχέση με τις διαδικασίες της άλλες χώρες. Τι θα μας συμβουλεύατε, τι θα λέγατε, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να υποστηρίξουμε αυτά τα έργα. Merci beaucoup. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τιέν. Κύριε Ροντρίγκης, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και συγχαρητήρια στους συντονιστές για τις παρουσιάσεις τους. Έχω δύο γενικές ερωτήσεις και δύο πιο ειδικέ για το διάδρομο της Μεσογείου. Οι γενικές μου ερωτήσεις είναι οι εξής. Ερώτηση πρώτη πώς βλέπετε να επηρεάσει η πρωτοβουλία του δρόμου του μεταξιού την χαρτογράφηση των διαδρόμων και πώς θα γίνει η διασύνδεση των διαδρόμων αυτών με το δρόμο του μεταξιού. Αν να σημείωσα σωστά, υπολογίστε γύρω στο 1 δισεκατομμύριο το κόστος ε, του διαδρόμου της Μεσογείου. Το, η σύραγγα Γερμανίας ε, Δανίας είναι 7,1 δις. Μήπως ε, έτσι διατρέχουμε τον κίνδυνο να έχουμε πρώτη, πρώτης και δεύτερης κλάσης ε, διαδρόμους. Γιατί σε μερικούς διαδρόμους γίνονται προσπάθεια μείωση του κόστους και επίσης η ανώτατη επιτρεπόμενη ταχύτητα είναι 180 χιλιόμετρα. Αν θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερες επενδύσει, θα είχαμε περισσότερες πλατφόρμες, οπότε θα είχαμε υψηλότερε προδιαγραφέ ε, εφάμιλε με του μεγαλύτερου διεθνεί διαδρόμου. Επίση, στην περίπτωση του διαδρόμου της Μεσογείου η, Ευρωπαϊκή, η Ισπανική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας ε, είπε ότι είναι σωστή η μετάδοση και θα μπορούσε να πιστοποιηθεί ώστε να φτάσουμε μέχρι τα 220 χιλιόμετρα την ώρα ταχύτητα. Βέβαια, η πιστοποίηση ε, δεν ε, επετεύχθη, δεν εδόθη. Η συντονίστρια συμφωνεί ότι οι δοκιμές ήταν κατάλληλες και τα αποτελέσματα έγκαιρα ώστε να ε, δοθεί η πιστοποίηση και πώς ε, δικαιολογείται ότι υπάρχουν κάποια τμήματα αυτών των διαδρόμων που περνάνε από άλλες ε, τρίτες οδούς. Ο κύριος Φλέγκο. Ευχαριστώ. Έχω μια σύντομη ερώτηση για την κυρία Ελίζα Γένσεν. Με το ψήφισμα του 2016 για τη βελτίωση της διασυνδεσιμότητας των υποδομών μεταφορών στη Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε τη σημασία του λιμανιού Ριέκα στην Κροατία στις ευρωπαϊκές μεταφορές και ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσει ώστε το λιμάνι της Ριέκα να συνδεθεί με το διάδρομο Βαλτικής Αδριατικής. Αυτός ο διάδρομος συνδέει τη σύγχρονη Αδριατική με τη Βαλτική και περνάει από την Αυστρία, τη Σλοβακία, τη Τσεχία και την Πολωνία. Στην διασύνδεση αυτή, στο διάδρομο αυτό, πότε αναμένεται η αναθεώρηση, η αξιολόγηση μάλλον του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών και θα λάβει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη συστάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να συμπεριλάβει και το λιμάνι της Ριέκα και να του δώσει αντίστοιχο καθεστώς εφάμιλο με αυτό ότι ε, στριέστης, τεριέστης της Βενετίας και άλλων ε, σημαντικών λιμανιών. Και έχουμε δύο ε, ευρωπαϊκούς διαδρόμους που θα, ή θα, μπορέσει να συνδεθεί και με άλλο διαδρομούς ή μόνο με το διάδρομο Βαλτικής Αδριατικής. Καλώς, ελήφθη το μήνυμα. Κυρία Τάλερ, ένα λεπτό μόνο. Ευχαριστώ πολύ αγαπητή Πρόεδρε θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος του συναδέλφου Τζουζέπε Μιλάτσο που κολλείεται, αλλά θέλει να κάνει ερώτηση. Γι' αυτό θα το γυρίσω στα αγγλικά, γιατί δυστυχώς στα ιταλικά δεν τα ομιλώ. Στην πολιτική των διευρωπαϊκών δικτύων η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει ε, να βελτιώσει το δίκτυο των υποδομών. Υπάρχουν όμως περιφερειακές ζώνες που παραμένουν εκτός των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων. Περιφέρειες όπως η Νότια Ιταλία, για παράδειγμα, έχουν ακόμα καθυστέρηση και στις υποδομές και στη σύνδεση που επηρεάζει αρνητικά την οικονομία και ε, την οικονομία χωρίς αποκλεισμούς, που είναι βασικός στόχος της πολιτικής των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Έχετε να μας δώσετε κάποια θετικά μηνύματα σχετικά ότι θα αλλάξει πορεία και αν ναι, προς ποια κατεύθυνση. θα μπορούσατε να μας το περιγράψετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Νόβακ. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ. Αναφέρατε δύο φορές ότι ε, διέρχονται δύο διαδρομοί από το κόπα στην Σλοβενία. Πολύ σημαντικό μέρος. Η Σλοβενία είναι χώρα ε, διέλευσης από ανατολάς προς και αντιστρόφως έχουμε χτίσει άριστους αυτοκινητοδρόμους απλά έχουν γεμίσει φορτηγά. Χρειαζόμαστε σιδεροδρόμους. Δυστυχώς Έχουμε την αίσθηση στη Σλοβενία ότι όλα πάνε υπερβολικά αργά. Και σας ρωτώ, θεωρείτε ότι η πρόοδος είναι αρκετή όσον αφορά τη συνεργασία με τη σλοβενική κυβέρνηση, όσον αφορά την υλοποίηση αυτών των σιδηροδρομικών διαδρόμων μέσω της Σλοβενίας και σε θέματα χρηματοδοτικά τα κονδύλια αυτά θα διατεθούν και στην στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Η Νάπολη και το Σαλέρνο είναι δύο περιοχές της ε, καμπανίας ε, ε, της Νότιας Ιταλίας, της επαρχίας, συγγνώμη, της Ιταλίας. Από την Νάπολη περνούν επιβάτες και εμπορεύματα σε τεράστιους αριθμούς και από το αεροδρόμιο και από το λιμάνι. Και εκεί υπάρχουν υποδομές ε, αυτής της διαδρομής ε, που συνδέει τη Μεσόγειο με την Σκανδιναβία. Στο λιμάνι του Σαλέρνο ε, θεωρείται ότι έχει στρατηγική περιφερειακή όμως ε, σημασία. το αεροδρόμιο του Σαλέρνο δεν λαμβάνεται υπόψη. Ερώτηση προς τον κύριο Κόξ. Δεν θεωρείται ότι θα πρέπει και αυτή η περιοχή να έχει ένα επιπλέον ή εναλλακτικό λιμάνι από αυτό της Νάπολης. Το λιμάνι και το αεροδρόμιο της Νάπολης λόγω του τουρισμού έχουν τεράστιες αφήξεις και αναχωρήσεις αφού επανεξετάζουμε τους ευρωπαϊκούς διαδρόμους θα μπορούσαμε να σκεφτούμε κάποια αναβάθμιση για το αεροδρόμιο και το λιμάνι του Σαλέρνο αφού έχουν στρατηγική σημασία τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο και ποια θα μπορούσε να είναι η εξέλιξη του, διαδρόμου Σκανδιναβίας Μεσογείου σε, ε, σε επίπεδο στρατηγικό και δομικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για όλες τις ερωτήσεις σας. Έχω και εγώ δύο ερωτήσεις και για ποιο λόγο να μην τις κάνω. Ε, αλλάζω ιδιότητα λοιπόν τώρα. Έχω ένα προβληματάκι γιατί ακούμε ότι οι διάδρομοι είναι για να γίνουν πιο ρευστά τα πράγματα στην Ευρώπη και να μπορεί κανείς πραγματικά να πηγαίνει από τη μια πρωτεύουσα στην άλλη. Έχω λοιπόν το εξής πρόβλημα. Μεταξύ σας μιλάτε καμιά φορά. Οι συντονιστές, συντονίζεστε, συνεννοείστε Μήπως θέλουν συντονιστεί και οι συντονιστές για το συντονισμό τους. Πώς είναι δυνατόν το 2019 να μην ε, πάω Παρίσι-Βερολίνο με ένα νυχτερινό τρένο, αν δεν θέλω να πάρω αεροπλάνο. Λέω, βλέπω τους Γερμανούς γιατί βλέπω ε, τα αιτήματα των ε, Γερμανών που θέλουν να ταξιδεύουν σε άλλες χώρες με τρένο και μάλιστα με νυχτερινά τρένα. Και δεν τα βρίσκω γιατί δεν υπάρχει νυχτερινό τρένο Παρίσι-Βερολίνο. Έχω πρόβλημα. Γιατί πρέπει να απαντήσω και για το κλίμα και για το χρήμα. Πρέπει κάτι να βρούμε και κοιτάμε το χάρτη και λες βρε παιδάκι μου δεν είναι δυνατόν να μπορεί κανείς ως Ευρωπαίος πολίτης να πηγαίνει από το ένα μέρος στο άλλο στην Ευρώπη με ε, μέσον που δεν ρηπαίνει ή λιπαίνει λιγότερο. Πόσο πιο ωραίο δεν θα ήταν να είναι το τρένο ε, προτεραιότητα. Μήπως θέλετε λοιπόν κανένα συντονιστή κι εσείς για να ταρακουνήσει λίγο τους ηγέτες και τους υπουργούς και αν δεν μπορούν να τους βοηθήσουμε για να συντονιστεί το δίκτυο και να μην έχουμε κάποιους μικρούς διαδρόμους. Πρώτη ερώτηση ήταν αυτή. Ερώτηση δεύτερη. Όσοι με γνωρίζουν, ξέρουν ότι έχω πρόβλημα με ένα μεγάλο έργο που λέγεται Λιόν Τωρίνο, η Σύρια γκάφτη. Πού βρισκόμαστε Μπορείτε να μας δώσετε κανένα ποσό για την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της σύρεγγας αυτής. Και ποιο είναι το κλάσμα που ήδη έχει δαπανηθεί. Για ποιο λόγο το λέω αυτό. Γιατί αν φτιάχνουμε σύραγγα, γιατί διάβασα όλες τις μελέτες και τα λοιπά, και τους υπέρ και τους κατά, ουσιαστικά το 2032 θα ολοκληρωθεί αυτό το έργο και τώρα είμαστε στο 2019. Εμένα δεν με πειράζει, εντάξει, εμπορευματικέ μεταφορέ, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το 2032. Ρωτάω, δεν νομίζω. Άρα, κάποια στιγμή δεν θα πρέπει οι διάδρομοι να έχουν ένα μεγάλο σχέδιο χρηματοδότησης για την ανανέωση του σιδηρομικού δικτύου και δεν είστε εσείς άραγε οι καλύτεροι σύμμαχοί μας και για τις επιβατικές και για τις εμπορευματικές μεταφορές. Εγώ νομίζω ναι. Μπορούμε να συνεργαστούμε. Και τελευταία μου ερώτηση είναι η εξής. Και θα επανέλθω και στην ερώτηση του κυρίου Ρικέ. Εσάς, σας ρώτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, όταν έκανε την πρόταση για τα smart, τα έξυπνα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Έχουμε πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Θα σας δώσω όχι πέντε λεπτά, τέσσερα στον καθένα για να μπορέσετε να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Et si on par vous, monsieur Patcox Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από εσά, κύριε Πατκόξ, να ακολουθήσουμε την αντίστροφη σειρά τώρα. Βεβαίω. Πολλέ ερωτήσει τέθηκαν. Θα διαλέξω μερικέ για να απαντήσουν και οι άλλοι συναδελφοί. Η κυρία Τάιλερ μίλησε για ειδικά γραφειοκρατικά εμπόδια. Υπάρχει μακροσκέλη κατάλογος τέτοιων. Για να σα δώσω ένα απλό παράδειγμα. Είναι σχεδόν αδύνατο από τα περιφερειακά και τα εθνικά σύνορα να περάσουμε, ιδιαίτερα στην περιοχή του Μπρένερο, να βρούμε συμφωνία για μια κοινή ταρίφα των διοδίων. Ε, μακάρι να μπορούσαμε να συντονιστούμε και να μα βοηθήσει σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο. Επίση, δεν μπορούμε να μιλήσουμε με του Αυστριακού για τα σχετικά χαμηλά, τις χαμηλούς φόρους, κατανάλωση φόρους κατανάλωσης που έχουν για τον δίζελ. Ενώ έχουμε 300 με 300-400 χιλιάδες φορτηγά που περνάνε από τον Μπρένερ μόνο και μόνο για να αγοράσουν φθηνότερα καύσιμα. Αυτό είναι επιλογή των Αυστριακών, δεν είναι ευρωπαϊκή επιρροή. Σκεφτείτε το. Επίση, χρειαζόμαστε περισσότερε επενδύσει στα δερματικά. Δεν έχουμε αρκετού δερματικού σταθμού, γιατί έχουμε 740 μέτρα μήκο ε, που θα είναι το στάνταρ ε, για το μήκο των σιδηροδρόμων, των, των τρένων. Ε, Επίση, ε, πώ θα Πώς θα τα λύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Είναι μακροσκελής ο κατάλογος των προσκομμάτων των γραφειοκρατικών. Για τα ορόσημα. Ολοκληρώσαμε 109 μέτρα, ε, χιλιόμετρα, συγγνώμη, ε, μέτρα σύραγγας. Δεν είναι δύσκολο. Έχουμε ακόμη 290 και ελπίζω θα το ολοκληρώσουμε στα τέλη του 2023 μέχρι το 2024. Αυτό θα ήταν σημαντικό ορόσημο και θα πρέπει να το εξοπλίσουμε μετά. Και αυτό είναι το βασικό θέμα. Θέλουμε ε, επιχειρησιακά, όχι απλώς να έχουμε ένα σύστημα διαφορετικό σύστημα σήμανσης στα διάφορα τμήματα του διαδρόμου, άλλο στην Αυστρία, άλλο στην Ιταλία. Θέλουμε ένα ενιαίο σύστημα από το Μόναχο στη Βερόνα. Και αυτό θα είναι δύσκολο να το επιτύχουμε. Θέλουμε μια ενιαία ευρωπαϊκή προσέγγιση, ευρωπαϊκό όραμα. Χωρίς ευρωπαϊκό όραμα καμία χρηματοδότηση. Και τι θα έλεγα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δύο μήνυματα. Καταρχήν, θα πρέπει να επιμένουμε σε όλα τα επιμέρους σχέδια και να έχουμε μια εφαρμοστική οδηγία για κάθε επιμέρους σχέδιο. Η, εφαρμοστική οδηγία ε, δίνει ορόσημα, υποχρεώνει σε ενημέρωση και εκθέσεις, υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν πιο στενά με το συντονιστό, ώστε να έχουμε έργο, να παράγουμε έργο και να έχουμε καταμετρήσιμα αποτελέσματα. Θα πρέπει κάθε τέτοιο μείζον σχέδιο να συνοδεύεται από οδηγία εφαρμογή. Επίση, απαλλαγή ε, από, τα καυσαέρια, από τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Σίγουρα ε, χρειαζόμαστε κάποιες σημαντικές ρηξικέλευθες αλλαγές, δραματικές. Αν θέλουμε ε, αλλαγές, δεν αρκούν κάποιες εμβαλωματικές λύσεις και διάμεσες αλλαγές, αλλά πραγματικά ρηξικέλευθες, επαναστατικές αλλαγές. Και τώρα για τις μεταφορές όσο μεγαλύτερη πιθανότητα να μεταβούμε στα ηλεκτρικά οχήματα, που είναι πραγματικά τεράστιο το δυναμικό, όσο περισσότερο θα έχουμε τέτοια μετάβαση, θα αυξηθεί το, η ζήτηση του ηλεκτρικού ρεύματο, που θα πρέπει να προέρχεται από ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, όχι από λιγνίτη και από άνθρακα ε, ή από πυρηνικά, που στη Γερμανία ε, περιορίζονται. Ε, θα έχουμε τεράστια ζήτηση ηλεκτρικού ρεύματος. Οπότε δεν μπορούμε να μιλούμε μόνο για τι μεταφορέ ε, και να τι βάλουμε σε ένα στεγανό. Θα πρέπει να το δούμε σε συνδυασμό με την ενέργεια. Και χρειαζόμαστε και ένα ψηφιακό σκέλο. Το θέμα των διευρωπαϊκών δικτύων, που είναι ενέργεια, μεταφορέ και ψηφιακά θέματα, θα πρέπει όλα αυτά να τα ε, εφοδιάσουμε με φιλοδοξία, με πυγμή και να ζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα συνδυάσει. Γιατί ο καθένα ξεχωριστά μπορεί να αποτύχει, αλλά από κοινού μπορεί να επιτύχουμε τι ρηξικέλευτε αλλαγέ που απαιτούνται. Επίσης, για το εφιέστημα των μεταφορών, και αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Την περασμένη εβδομάδα αφιέρωσα πολλές μέρες στη Στοκχόλμη και συμμετείχα σε πολλές παρουσιάσεις, σε διασκέψεις, ανάλυση πολιτικής στη Σουηδία και Τι θα γίνει με αυτά τα σκούτερ τα ηλεκτρικά στις πόλεις, με ρώτησαν, θα χρειάζεται ρύθμιση. Στη Στοχόλμη δεν υπάρχει κανονιστική ρύθμιση. Αλλά υπάρχει ψηφιακό ε, έλεγχο ε, τη ταχύτητα. Δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 6 χιλιόμετρα την ώρα. Με ένα τέτοιο ψηφιακό έλεγχο μπορούμε να επιτύχουμε το αποτέλεσμα. Όλε αυτέ είναι πολύ καλέ ιδέε για αυτά τα ηλεκτρικά πατίνια και σίγουρα Θέλουμε έξυπνες λύσεις και μπορούμε να διδαχθούμε από ανθρώπους που είναι και ξυπνότεροι από μας. Ευχαριστώ. Η κυρία Ράντι Τσόβα για τέσσερα λεπτά επίσης. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας, τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω αυτά που μπορώ να απαντήσω τι έχω να προτείνω στην ε, Ευρωπαϊκή Επίτροπο ή την Ευρωπαϊκή Επίτροπο. Οι κυβερνήσεις στα χέρια τους πάντα έχουν κάποιο είδου πιθανούς κανονισμούς και πάντα οθούν τις κοινωνίες προς, για παράδειγμα, πιο περιβαλλοντικές, περιβαλλοντικά φιλικές προσεγγίσεις. Για να έχουμε λοιπόν ε, μεγαλύτερη απαλλαγή από ανθρώπινε εκπομπέ και το λέμε σοβαρά αν θέλουμε πραγματικά μια πράσινη Ευρώπη πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να υποστηρίξουμε τις ιδεοδρομικές μεταφορές και να είναι ανταγωνιστικές με τις μεταφορές ε, μέσω αυτοκινητοδρόμου. Με άλλα λόγια, αν συγκρίνουμε, όταν συγκρίνουμε ταχύτητα, τιμή και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, Το καλύτερο είναι όταν η ταχύτητα είναι ικανοποιητική, η τιμή είναι χαμηλότερη και η περιβαλλοντική επίδραση καλύτερη. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να συζητήσει με τις κυβερνήσεις κομισιών και πιστεύω θα συζητήσουμε με τις εθνικές κυβερνήσεις για το πώς μπορούμε να αλλάξουμε την προτεραιότητα που έχουν οι αυτοκινητόδρομοι λόγω τιμής και ταχύτητας κυρίως. Ώστε να προωθήσουμε περισσότερο τους σιδηροδρόμους, δημιουργώντας σιδηροδρόμους πιο ε, ικανοποιητικούς από τους αυτοκινητοδρόμους, διότι τώρα είναι ακριβή, είναι αργή και οι συνδέσεις δεν είναι ακόμα έτοιμες. Από τη δική μου άποψη ε, αυτές είναι οι προτεραιότητες. Κάτι δεύτερο. Δεν μπορούμε παρά να δώσουμε μερικές συμβουλές σε κυβερνήσεις, τίποτα άλλο. Να τους δώσουμε κάποια θετικά κίνητρα, να κινητοποιηθούν περισσότερο ε, όσον αφορά τις συνδέσεις των διαδρόμων. Διότι όπως γνωρίζετε δεν είναι μόνο θέμα αρμοδιοτήτων αλλά και οικονομικών. Το 50% της συγχρηματοδότησης προέρχεται από ευρωπαϊκές πηγές, αλλά ένα άλλο κομμάτι είναι αρμοδιότητα εθνικών κυβερνήσεων. Αν οι κυβερνήσει δεν συμβάλλουν και δεν καταβάλουν προσπάθειες, δεν υπάρχει κανένα τρόπο να φτιαχτεί ένα διάδρομο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μιλήσατε για κάποιες μη ανεπτυγμένε συνδέσεις στην Νότια Ιταλία, σε άλλες περιοχές. Ναι, το ξέρω. Αλλά είναι αρμοδιότητες και ευθύνε των τοπικών και περιφερειακών και εθνικών κυβερνήσεων. Ζήτα συγγνώμη η ομιλήτρια. Δεν είναι ούτε καθήκον ούτε σκοπός του διαδρόμου. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε και αυτό ισχύει για τη Γαλλία και πολλές άλλες χώρες είναι να υποστηρίξουμε ανοιχτά τους ε, οδούς πρόσβασης στους διαδρόμους. Δηλαδή όλο και περισσότερες περιφέρειες να εμπλακούν ώστε να είναι πιο γνωστός ο διάδρομος, ε, να, είναι πιο αποτελεσματικός. Αυτό μπορούμε να κάνουμε και θεωρητικά δεν υπάρχουν όρια στη χρήση ευρωπαϊκών πόρων για την οικοδόμηση οδών πρόσβασης βήμα προς βήμα όταν αυτό έχει νόημα ή τουλάχιστον να συζητηθεί αυτό. Αν λοιπόν η Γαλλία αναρωτιέται πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει πραγματικά διαδρόμους ή όχι, αν το διερωτώνται και άλλες χώρες, αυτό εξαρτάται από τις οδούς πρόσβασης. Αλλά οι πολιτικοί θέλουν να το κάνουν, διότι χωρίς αυτά δεν έχει νόημα το όλο εγχείρημα. Και τέλος, καταλαβαίνω κυρία Πρόεδρε το, η στάση σας. Ναι, κάποιοι άνθρωποι είναι ιδιαίτερα επικριτικοί όσον αφορά τη σειρά γκαλιών το Και το αντίθετο υπάρχει, κάποιοι έντονοι υποστηρικτές. Αλλιώς δεν θα είχαμε φτάσει σε τέτοια φάση ε, κατασκευής του διαδρόμου. Εγώ για ένα έτος ε, ε, που βρίσκομαι στη θέση που βρίσκομαι έχω μελετήσει το ιστορικό της αντιπαράθεση και των συζητήσεων και θυμάμαι ένα σημαντικό πράγμα. Υπάρχει απόφαση της κυβέρνησης και στη Γαλλία και στην Ιταλία κοινοβουλευτική απόφαση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Υπάρχει συμφωνία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι εγώ ως Ευρωπαία Συντονίστρια δεν έχω κανένα δικαίωμα. να αμφισβητήσω αποφάσεις εκπροσώπων της κυβέρνησης, των κυβερνήσεων. Κανένα δικαίωμα. Η θέση μου λοιπόν είναι ότι υποχρεούμε να λάβω υπόψη μου τις αποφάσεις αυτές να κάνω ό,τι μπορώ καλύτερο για να προωθήσω την υλοποίηση ήδη ε, συμφωνημένων έργων. και χρημάτων που έχουν κατα... Ε, εκχωρηθεί για αυτά τα έργα. Τέλος, όσον αφορά το μερίδιο των χρημάτων από το συνολικό προπολογισμό για την Μεσογειακό Διάδρομο για το Λιόν Τωρίνο, δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Αυτό που με ρωτάτε είναι ο συνολικό σχεδιασμένος προπολογισμό που είναι 8,6 δις ή τα επιμέρους μέρη κατασκευής του διαδρόμου από διάφορες ε, περιόδους ε, δημοσιονομικές διαφέρουν. Αλλά αυτό που θα ήθελα να τονίσω και να μην το ξεχνάμε Πού να ξέρει κανείς, μπορεί να πλησιάσει και άλλη οικονομική κρίση. Εγώ στην τελευταία κρίση το 2008-9-10 θυμάμαι ότι τα πάντα άλλαξαν. Ήμουν πρωθυπουργό και όλα άλλαξαν από τη μια μέρα στην άλλη. Οπότε ποιο ξέρει τι μορφή θα έχει ο προπολογισμό. Από εσά εξαρτάται. Εσεί θα αποφασίσετε τον προπολογισμό. Το Συμβούλιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποφασίσει τον προπολογισμό. Επιπλέον, αν η κρίση όπως ελπίζω δεν είναι τόσο βαθιά όλα τα πράγματα θα αλλάξουν σε κάποιο βαθμό και θα ξανασυζητήσουμε τι θα κάνουμε με τους διαδρόμους είμαι βέβαιη ότι όπως τα πράγματα άλλαξαν το 2008, 2009, 2010. εντελώς άλλαξαν τελείως ευχαριστώ πολύ Merci pour vos Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις. Θα δώσω το λόγο τώρα στον Πάβελ. Πάβελ. Ευχαριστώ. Ε, στις πιο ειδικέ ερωτήσεις για το Ρήνο, πρώτον, φυσικά γνωρίζουμε τα προβλήματα στο Ρήνο, ιδιαίτερα με την ξηρασία που πέφτει στάθμη. Και ξέρετε ότι υπάρχει ένα σχέδιο ε, που έχει ε, προτείνει για τις εσωτερικές προωτές οδούς το Υπουργείο Μεταφορών ανάμεσα στο, στο και ε, μια πόλη πιο κάτω έχουν προτείνει να, να βαθύνουν το ρήνο. Είναι πολύ ακριβές αυτές οι εργασίες όμως για τις υποδομές. Και ρωτήσατε για τη σιδεοδρομική γραμμή Στουτγάρδη-Ούλμ είναι της κυρίας Κάρλα Πέις που θα έρθει κάποια στιγμή στο μέλλον που είναι η συντονίστρια για τα εναλλακτικά καύσιμα που ρώτησε κάποιος συνάδελφος βεβαίως ε, υπάρχει ένα ειδικό έργο εκεί ε, της ΙΝΕΑ για τη χρηματοδότηση εναλλακτικών καυσίμων και το ENTMS είναι η διευκόλυνση ε, Blaming αυτή ε, και θα συνεχιστεί. Έγινε μια γενική ερώτηση για το οικονομικό όφελος και πολλοί ρωτήσατε. Ξέρετε, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα πάντα στις υποδομές. Δεν υπάρχει ορατότητα ε, των θετικών εξωτερικών δράσεων. Ε, ε, είναι δύσκολο. Ε, περιμένουμε, ας πούμε, να γίνει ένας δρόμος, ένας σιδηρόδρομος, ένας αυτοκινητόδρομος, αλλά δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι θα υπάρχει οικονομικό όφελος. Υπάρχει όμως το αποτέλεσμα της μη ολοκλήρωσης του έργου. Και τα αποτελέσματα των μελετών τι δείχνουν, ότι αν δεν ολοκληρώσουμε τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, όπως έχει προβλεφτεί μέχρι το 2030, θα χάσουμε 1,6% του ΕΠ. Αυτό είναι βέβαια με βάση κάποιες παραδοχές που κάνουν οι οικονομολόγοι, αλλά ε, πρέπει να το συζητήσουμε. Η κυρία Γκαρσία Μουνιώθ ρώτησε για τις τράπεζες και πώς μπορούμε να κινητοποιήσουμε περισσότερο το ιδιωτικό κεφάλαιο. Δύσκολο είναι αυτό, γιατί θα πρέπει να έχουμε και έσοδα ε, και θα πρέπει να είναι επωφελές αυτό το έργο και να αποδίδει για τις υποδομές. Ε, πώς θα γίνει αυτό, πώς θα το αποδείξουμε ότι αποδίδει, γιατί για τις περισσότερες υποδομές ε, θεωρούνται δημόσιο αγαθό. Ε, στους αυτοκινητοδρόμους ε, μπορούμε να έχουμε τα ομόλογα έργου, όπως είναι ο αυτοκινητόδρομος ε11 ε, ή για κάποια ποτάμια, αλλά για σας είναι πολύ σημαντικό το εξής ερώτημα για σας τους βουλευτές. Πώς θα βρεθεί η ισορροπία ανάμεσα στις διάφορες μεταφορές, μέσα μεταφοράς. Θέλετε να φύγετε από το αυτοκινητόδρομο να πάτε στο σιδηρόδρομο. Και μίλησε ε, και για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, ο Πατ Κόκ, σε σχέση με το αυτοκίνητο ε, οι Ελβετοί ε, έκαναν παραμετροποίηση. Δηλαδή είναι πιο φτηνός ο σιδηρόδρομος ως μέσο μεταφοράς και πιο ακριβό το αυτοκίνητο. Μόνο έτσι γίνεται. Αυτό λέγεται εσωτερήκευση του εξωτερικού κόστους. Αυτό θα μπορούσε να γίνει, ε, αν όχι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωση, σε επίπεδο κρατών μελών. Αλλιώς δεν υπάρχουν πάρα πολλέ ελπίδες. Έγιναν και δύο ερωτήσεις. ως προς το... γιατί έχουμε ξεχάσει τις πιο απομακρυσμένες περιφέρειες ή τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες, γιατί εδώ μιλάμε για το κεντρικό δίκτυο. Γιατί από την πλευρά της ανταγωνιστικότητας το κεντρικό δίκτυο αποδίδει περισσότερο. Δεν σημαίνει όμως ότι, δεν θα πρέπει, ε, ότι θα πρέπει να ξεχάσουμε μάλλον τις άλλες περιφέρειες. Αλλά αυτό είναι στα κράτη των κρατών μελών. Γιατί εδώ τα ωφέλη τα οποία μας απασχολούν ε, ε, έχουμε βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχει να κάνει αυτό με την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Και όταν έχουμε διασυνοριακή υποδομή, γι' αυτό είναι και ο διάδρομος, όταν ε, αφαιρέσει τη συμφόρηση από ένα κράτος μέλο θα υποφεληθεί και κάποιο άλλο και το σύνολο του διαδρόμου. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε αυτή τη δομή για τη διακυβέρνηση. Και ρώτησε κάτι και η Καρίμα, αν μιλάμε μεταξύ μας, πολύ καλή ερώτηση. Βεβαίως, έχουμε το κολέγιο των συντονιστών, κάνουμε πολλά πράγματα μαζί, προτείνουμε καλές λύσεις και μαζί με τη Γενική Διεύθυνση μου, προτείνουμε ε, πάντα να προχωρούμε. Και η τελευταία ερώτηση είχε να κάνει αυτό που ρώτησε ο κύριος Ντάνιελσον, ε, τι συμβουλή θα δώσουμε στη νέα Επίτροπο. Να είναι πιο ορατή, να ζητάει περισσότερα χρήματα, να βάλει περισσότερους όρους και να συνεργάζεται με τους συντονιστές. Και ένα τελευταίο σχόλιο που είναι μια κινέζικη παροιμία. Αν θέλεις κάτι να, ε, αν θες να αναπτυχθείς, ε, ανάπτυξε τις υποδομές σου. Σας ευχαριστώ. Και η τελευταία μας συντονίστρια, κυρία Γένσεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα περιοριστώ σε τρία θέματα. Το πρώτο αφορά την ερώτηση του κυρίου Ντάνιελσον. Τι θα πούμε στον αρμόδιο επίτροπο. Όπως και ο Πάβελ, θα συνιστούσα στην επίτροπο να κάνει αυτή την παρουσία της και να ζητήσει περισσότερα κονδύλια ε, για να ολοκληρωθούν αυτά τα σχέδια μέχρι το 2030. Οπότε θα πρέπει να προβληθεί περισσότερο η αρμόδια επίτροπος και να ζητήσει τέτοια κονδύλια και να τα αυξήσει γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε πιο οικολογικές τις μεταφορές και να έχουμε τη μετάβαση από το δικό δίκτυο στο σιδηροδρομικό, αν δεν χρηματοδοτήσει τα προγράμματα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι απολύτω απαραίτητη χρηματοδότηση ευρωπαϊκή. Αυτή είναι η πρώτη συμβουλή που θα έδινα στην Επιτροπή. Υπάρχει και το θέμα των έξυπνων διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Τα κράτη-μέλη έχουν εκδηλώσει ζωηρό ενδιαφέρον, τουλάχιστον ε, όσα επισκέφθηκα εγώ. Πάντως, ε, θα βοηθούσατε τα κράτη να γίνουν πιο αποτελεσματικά προτείνοντας σημαντικά σχέδια και γι' αυτό θα πρέπει να μειωθεί ή να πλουσευτεί η γραφειοκρατία και διασυνοριακά να μειωθεί η γραφειοκρατία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άλλη συμβουλή. Πολλοί ρώτησαν το θέμα της εξάπλωσης των διαδρόμων, της επέκτασης των διαδρόμων. Γιατί ο ποταμός Όντερ δεν ε, είναι τμήμα του διαδρόμου. Ο κύριος Φλέγκο μίλησε για το λιμάνι Ριέκα στην Κροατία. Ε, επίσης και κάποιοι από τη Σουηδία ρώτησαν γιατί δεν μπήκε και η Σουηδία. Ε, γιατί υπάρχουν ε, πολωνικά, σουηδικά λιμάνια που συνδέονται με τα πολωνικά. Και γιατί δεν μπαίνουν τα σουηδικά λιμάνια σε αυτό το διάδρομο Βαλτικής Αδριατικής. Υπάρχει όμω κάποιο λόγο γι' αυτό. Υπάρχει... Έχει αξία αυτό το σχέδιο των διαδρόμων. Γι' αυτό και υπάρχει πιο ζωηρό ενδιαφέρον για συμμετοχή στου διαδρόμου. Θα πρέπει λοιπόν ε, να γίνει η αξιολόγηση και αναθεώρηση των διευρωπαϊκών δικτύων που αναμένεται για το 2023, αλλά ίσω ε, μετατοπιστεί το νωρίτερο από την Επίτροπο, που θα ήταν ε, πολύ σωστό, γιατί η νέα δημοσιονομική περίοδος, το νέο πολιτή δημοσιονομικό πλαίσιο θα αρχίσει από το 2021, οπότε έχει νόημα να γίνει νωρίτερα η αξιολόγηση των διευρωπαϊκών δικτύων και να μην περιμένουμε το 2023. Θα πρέπει ε, να δούμε μετά την αξιολόγηση πώς θα διαμορφωθούν στο μέλλον τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Και το βλέπω αυτό κυρίως με τις νέες χώρες που προσέκρουσαν ε, ε στο πρόβλημα να εγκρίνουν πολλά σχέδια, αλλά να μην έχουν χρηματοδότηση. Επίσης, το τελευταίο ζήτημα είναι το πρασίνισμα που λέμε. Την πρόσδεση πιο φιλοπεριβαλλοντικού χαρακτήρα, οικολογικού χαρακτήρα στα σχέδια και στις μεταφορές. Στις διαφάνειές μου είχα πολλά αεροδρόμια και φυσικά υπάρχουν τα αεροδρόμια και η αποτελεσματικότητα των αεροδρομίων μπορεί να βελτιωθεί. Αν βελτιωθούν οι διασυνδέσεις, δεν χρειαζόμαστε περισσότερα αεροδρόμια, αλλά να αξιοποιήσουμε τα υπάρχοντα αεροδρόμια. Αλλά και πάλι θα πρέπει να μεριμνήσουμε επαρκείς σιδηροδρομικές μεταφορές και κατάλληλο σιδηροδρομικό δίκτυο. Στο δικό μου διάδρομο, δύο χώρες ε, ενεργοποιούνται ιδιαίτερα στο τομέα αυτό. Η Τσεχία, που έχει πολύ φτηνέ και αποτελεσματικέ σιδηροδρομικές μεταφορές με έντονο ανταγωνισμό, που σημαίνει ότι ο κόσμος προτιμά το σιδηρόδρομο από το ιοταχή και επίσης και η Αυστρία διαπιστώνει ότι προωθεί τι σιδηροδρομικές μεταφορές. Θέλουμε λοιπόν περισσότερη εστίαση των κρατών μελών στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Και θα ήθελα να προσθέσω αυτά που είπε ο Πατ Κόξ για τα ηλεκτρικά οχήματα και ε, να καταστήσουμε πιο οικολογικές τις οδικές μεταφορές, χρησιμοποιώντας ευφυείς e συστήματα μεταφορών. Εκεί υπάρχει τεράστιο δυναμικό για πιο φιλοπεριβαλλοντικές μεταφορές, ιδιαίτερα στις οδικές μεταφορές. Και αυτό το θέμα σίγουρα θα μας απασχολήσει ιδιαίτερος στο εγγύς μέλλον. Σας ευχαριστούμε κυρία Γέρνησεν, ευχαριστώ όλους τους συντονιστές για την παρουσίαση. Είδαμε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλά κονδύλια, δεν ξέρουμε ακριβώ πώ χρησιμοποιούνται και αυτό δυσκολεύει τα πράγματα. Το λέω καθαρότατα. Μα λέτε θέλουμε στόχου. Ο στόχο έχει αναφερθεί δύο φορέ από την Πρόεδρο τη ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε έναν στόχο μείωση κατά 55% του διοξιδίου του άνθρακα. 55% λιγότερο διοξιδίου του άνθρακα μέχρι το 2030, δηλαδή ουσιαστικά αύριο. Αντιλαμβάνεστε τι μετασχηματισμούς απαιτεί αυτό το μείον 55%. Τι τα έργα που έχουν υψηλές εκπομπές πρέπει να τα απορρίπτουμε, να βρίσκουμε εναλλακτικέ. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να μαχηθούμε για πραγματικά έργα, αλλά να αντιστοιχούν στους στόχους που έχουμε θέσει μαζί. Οι μεταφορές πρέπει και αυτές να πραγματοποιήσουν τη μετάβαση αυτή, τη μεταβολή. Και, και εκεί κερδίζουμε όλοι, διότι όταν φτιάχνουμε υποδομές ξέρετε, θα μα ε, ζητήσουν ευθύνε σε 20 χρόνια. Εμεί θα είμαστε οι αρμόδιοι για τις ε, υπεύθυνοι. Δεν είμαστε κατά τη πρόοδου, Βίκτορ, γιατί με κοιτάτε. Η ψηφιοποίηση θα παραμείνει στο επίκεντρο, αλλά δεν μπορούμε πια να κάνουμε τα πράγματα όπως στο παρελθόν. Είναι αδύνατον. Το δεύτερο που μου φαίνεται πολύ σημαντικό Και εγώ δεν έλαβα απάντηση γιατί δεν δόθηκαν απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα που ακούσαμε. Δεν ξέρουμε ποια είναι η θέση σας για το έξυπνα διευρωπαϊκά δίκτυα. Ε, αυτά που είπε ο κ. Φλεγκό προηγουμένω είμαστε απαντήσεις. Δεν λάβαμε όλες τις απαντήσεις. Σας καλώ λοιπόν να γράψετε στους συντονιστές μας ώστε να λάβετε απαντήσεις. Το τρίτο είναι ότι πρέπει να θέσουμε στόχους. Έχουμε πέντε χρόνια για να επιτύχουμε την συνδεσιμότητα όλων των κρατών μελών. Γιατί, διότι ο κόσμος χρειάζεται κίνηση. Αν μπορέσουμε να ομαλοποιήσουμε λοιπόν τις μεταφορές, η δράση πρέπει να είναι τώρα, όχι σε 10 χρόνια. Τώρα πρέπει να αναλάβουμε δράση. Τώρα πρέπει να ξεκινήσουμε τα σχετικά έργα. Αλλά όπως είπατε, σε ανθρώπινη κλίμακα, να χαρακτηρίζονται από εγκύτητα για να ξαναδώσουμε ζωή στην τοπική διάσταση. Αυτό είναι το μέλλον της κινητικότητας. Ευχαριστούμε για τις παρουσιάσεις σας. Πέρασε η ώρα γρήγορα και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Τους άλλως δεν είμαστε μακριά και ελπίζω ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα. Όλες οι ερωτήσεις λοιπόν που θεωρείτε ότι δεν απαντήθηκαν στείλτε τες απευθείας στους συντονιστές μας ε, τους οποίους ευχαριστώ και τα λέμε σύντομα. Και εμείς θα συνεχίσουμε φυσικά. Συνεχίζουμε, μην ξεχνιόμαστε αγαπητοί συνάδελφοι. Στην αρχή της κοινοβουλευτικής περίοδου κάλεσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας παρουσιάσει έτσι γενικώ τι θα κάνει για τις διεθνείς συμφωνίες ε, στις αερομεταφορές και ποιους στόχους έχετε γενικά. Όπως γνωρίζετε υπάρχουν διάφορες συμφωνίες αεροπλοείας ε, ορισμένες διέπουν τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες, ενώ κάποιες άλλες την ε, ασφάλεια στην εναέρια κυκλοφορία. Και έχουμε και με τη συνθήκη της Λισαβόνας ενισχυμένες ε, αρμοδιότητες και εξουσίες του Κοινοβουλίου σημαντικά, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει κατά τον νόμο να ενημερώνει το Κοινοβούλιο καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάποιες τρίτης χώρας, έτσι ώστε να μπορούν να τεθούν σε ισχύ και χρειάζεται ρητή έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όλα αυτά λοιπόν για τις διαπραγματεύσεις κανονικά είναι διαβαθμισμένα που σημαίνει ότι είναι λίγοι εκείνοι που έχουν πρόσβαση. Παρ' όλα αυτά, συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η σημερινή συνεδρίαση να είναι κατ' εξαίρεση δημόσια έτσι ώστε να μπορέσουν ε, όσο γίνεται περισσότεροι να υποφεληθούν και να απαντήσει πάνω κάτω δημοσίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σε κάποιες ερωτήσεις. Ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Κύριε Ερμέζο Κώστα. Ça va comme ça? Super. En ε, Καλά τα είπα στα Ισπανικά. Έχετε το λόγο για ένα τεταρτάκι, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, ε, Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους αυτό που θέλω να κάνω σήμερα να σας δώσω πολύ σύντομη επισκόπηση το, όσων κάνουμε ε, στις εξωτερικές συμφωνίες για την αεροπλοεία. Έχουμε προετοιμάσει μια σύντομη παρουσίαση. Να αρχίσω ευθύ εξ αρχής λέγοντας ότι καθ' όλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ενημερώνεται πλήρως το Κοινοβούλιο για τα τεκτενόματα, έχετε πρόσβαση στα διάφορα έγγραφα και χαιρόμαστε που έχουμε την ευκαιρία να έρθουμε σήμερα να σας ενημερώσουμε και να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας σε ό,τι αφορά τις αεροπορικές συμφωνίες έχουμε δύο μεγάλες ενότητες, αν μπορώ να το πω έτσι. Το ένα είναι οι συνολικές ε, συμφωνίες όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύεται ε, δυνατότητα, ε, δικαιώματα κυκλοφορίας, να πετάμε σε τρίτες χώρες δηλαδή, και άλλες συμφωνίες που έχουν να κάνουν σε μια βασική εταιρική σχέση. Έχουμε μια συμφωνία για δικαιώματα μεταφορών ε, αλλά ασφάλεια, ενεργική και παθητική, ε, θεμητό ανταγωνισμό και αυτές οι συμφωνίες έρχονται να αντικαταστήσουν τις συμφωνίες που έχουν διμερώς τα κράτη-μέλη. Γιατί ξέρετε ότι σήμερα εξακολουθούν τα κράτη-μέλη διμερώς να διαπραγματεύονται και μόνο όταν έχει εντολή Ευρωπαϊκή Ένωση να διαπραγματευτεί μια διεθνή συμφωνία. Αυτό γίνεται και για να γίνει αυτό χρειάζεται ομοφωνία. Πρέπει να συμφωνήσουν όλα τα κράτη-μέλη. Υπό την έννοια αυτή σήμερα λοιπόν έχουμε εννέα ε, συμφωνίες ε, ισχύ και διαπραγματευόμαστε άλλες οκτώ. Και θα έρθω τώρα στις λεπτομέρειες. Επίσης έχουμε και άλλες συμφωνίες που μπορεί να είναι λίγο πιο δύσκολο να κατανοηθούν. Τις ε, ονομάζουμε οριζόντιες εγκάρχες συμφωνίες. Ε, τι στόχουν αυτές να εξασφαλίσουν ότι οι διμερείς συμφωνίες που έχουν με τρίτες χώρες τα κράτη-μέλη σέβονται απολύτως το κοινοτικό δίκαιο. Γιατί όπως μπορεί να γνωρίζετε, ε, οι συμφωνίες που έχουν τα κράτη-μέλη διατυπώνονται με τέτοιο τρόπο που ε, να εποφελούνται από τη συμφωνία μόνο οι αερομεταφορείς ε, της χώρας αυτής. Ας πούμε, Ισπανία, Βραζιλία, εποφελούνται μόνο οι ισπανικές εταιρείες. Το 2002 υπήρξε απόφαση του δικαστηρίου για το κατά πόσο αυτό συνάδει με το ευρωπαϊκό δίκαιο και εμείς καλούμαστε να το κάνουμε αυτό. Πώς γίνεται αυτό. Είτε η ίδια η χώρα μέλος επαναδιαπραγματεύεται τη συμφωνία με την τρίτη χώρα ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξ ονόματος και των 28 με μία μόνο κονδυλιά εναρμονίζει με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο όλες αυτές τις συμφωνίες των κρατών μελών. Αυτές είναι οι οριζόντιες. Και μετά έχουμε και τις συνολικές, είναι, ε, καθολικές, comprehensive. Βλέπετε εδώ ένα χάρτη παγκόσμιο που, για τις συμφωνίες που έχουν ήδη υπογραφεί και εφαρμόζονται. Τα πράσινα είναι Καναδά, Ηνωμένε Πολιτείε, Ισραήλ, η Ορδανία, Μαρόκο, Μολδαβία και Δυτικά Βαλκάνια και Αυτές είναι οι συμφωνίες που εφαρμόζονται ήδη. Έχουμε κάποιες συμφωνίες όπου έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις αλλά δεν έχουν ακόμα υπογραφεί. Αυτές ε, λοιπόν έχουν τελειώσει αλλά δεν έχουν υπογραφεί άρα και δεν μπορούν ακόμα να εφαρμόζονται. Αρμενία, Κατάρ, Ισία, Ουκρανία είναι αυτές οι συμφωνίες. Για ποιο λόγο δεν μπορούμε να τις υπογράψουμε. Θα γνωρίζετε ήδη ότι έχουμε πρόβλημα με ε, τον ορισμό της επικράτειας λόγω του αεροδρομίου στο Γιβραλτάρ. Αυτό δεν έχει λυθεί ακόμα. Ελπίζουμε να λυθεί, αλλά προς το παρόν δεν εφαρμόζονται παρόλο που έχουν τελειώσει οι διαπραγματεύσεις. Και μετά έχουμε τρέχουσες διαπραγματεύσεις και θα επανέλθω σε συνέχεια. Εδώ είναι το κόκκινο. Ε, ε, βλέπετε και τις ημερομηνίε πότε έχουμε υπογράψει με την ε, Ουκρανία, Αρμενία, την και Κατάρ. Είπαμε έχουμε μονογράψει τη συμφωνία που σημαίνει ότι τελειώνουν διαπραγματεύσεις αλλά δεν έχουν ακόμα υπογραφεί άρα και δεν εφαρμόζονται. Και συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με κάποιες χώρες. ΑΣΕΑΝ, ε, Νότια Ανατολική Ασία που είναι 10 χώρες εκεί, Βιετνάμ, Ταϊλάνδη, Ινδονησία, Μαλαισία, Φιλιππίνες κλπ. Όλες μαζί, ΑΣΕΑΝ. Είναι διαπεριφερειακή αυτή η συμφωνία, πάρα πολύ σημαντική και περίπου έχουμε τελειώσει τις διαπραγματεύσεις. Ήμασταν ε, το Νοέμβριο στο τελευταίο γύρο, αλλά άλλαξε η κυβέρνηση σε μία από τις χώρες ΑΣΕΑΝ, στη Μαλαισία, που ζήτησαν περισσότερο χρόνο για να μελετήσουν τη συμφωνία και αυτές οι εσωτερικές διαβουλεύσεις η Μαλαισία ε, τραβάνε σε μάκρους περισσότερο από όσο ε, υπολογίζαμε, γι' αυτό και δεν έχουν ολοκληρωθεί τυπικά και επίσημα οι διαπραγματεύσεις και ελπίζουμε αυτό να γίνει προσεχώς. Επίσης συνεχίζονται με το Αζερβαϊτζάν οι συνομιλίες, ήταν μικρή πρόοδος ε, διότι υπήρχαν κάποια ζητήματα. Ε, το φθινόπωρο έχουμε τον επόμενο γύρο, ακόμα δεν ξέρουμε πότε τις ημερομηνίε και θα θέλαμε τέλη του έτους να ολοκληρώσουμε. Με την Τουρκία επίσης έχουμε εντολή να διαπραγματευτούμε. Κάναμε διάφορους γύρους, αλλά όπως ίσως γνωρίζετε το Συμβούλιο τον Ιούλιο αποφάσισε να μάλλον να διακοπούν, να ανασταλούν αυτέ οι διαπραγματεύσει λόγω τη γενικότερη πολιτική κατάσταση, Ένα από τα μέτρα που έλαβε το Συμβούλιο ήταν να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διακόψει ε, τις διαπραγματεύσεις Και η τελευταία ε, ε, συμφωνία που διαπραγματευόμαστε είναι με τον ΟΜΑΝ. Αρχίσαμε στι αρχέ του 19. Πηγαίνουν πολύ καλά διαπραγματεύσει. Ήδη έχουμε καταλήξει σε συμφωνία με το Κατάρ και αυτό διευκολύνει τα πράγματα. Και έχουμε τώρα το Νοέμβρη ένα νέο γύρο και ελπίζουμε να μπορέσουμε να επιτύχουμε μεγάλη πρόοδο σε όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις. Θα ήθελα επ' ευκαιρία τώρα να σας πω δύο λόγια ε, για τις ωφέλειες που έχουμε από τις Ευρωπαϊκές Συμφωνίες σε σχέση με τις διμερείς. Μετά την εφαρμογή της συμφωνίας έχουμε αύξηση σε αριθμό ε, επιβατών, ε, σε δρομολόγια με πόλεις που δεν συμμετείχαν και επίσης μειώθηκαν οι τιμές των εισιτηρίων. Ας πούμε, τις Ηνωμένε Πολιτείε έχουν αυξηθεί κατά 20% ο αριθμός των επιβατών. Είναι δύο όριμες αγορές, άρα δεν αναπτύσσονται πάρα πολύ όπως θα δείτε αλλού. Παρ' όλα αυτά έχουμε περισσότερα δρομολόγια ε, σε πόλεις που δεν υπήρχαν στο παρελθόν και 27% κατά μέσο όρο έχει μειωθεί το κόστος ε, του εισιτηρίου. Με τα Δυτικά Βαλκάνια, αντίστοιχα, για να σας πω ακόμα καλύτερα, ακόμα μεγαλύτερη αύξηση σε επιβάτες, ε, περισσότερες πόλεις, συν 125 διάδες πόλεων σε σύγκριση με το 2006 το ίδιο με το Μαρόκο, ε, περισσότεροι επιβάτες, περισσότερες πόλεις που συνδέονται και μείωση στο, ε, στη μέση των εισιτήριων. Ε, αντίστοιχα ισχύουν και για το Ισραήλ, είναι παρόμοια η κατάσταση. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι οι ευρωπαϊκές συμφωνίες φέρουν σημαντικά ωφέλη στους διάφορους ενεχόμενους. Από την άλλη, ε, αυτό ε, ε, ενδιαφέρει και το Κοινοβούλιο, είναι μακρά η διαδικασία κύρωσης, γιατί είναι εγώμενες μεικτές συμφωνίες. Τι σημαίνει αυτό. Θα πρέπει, είναι μέρη και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κρατη Άρα πρέπει να κυρωθούν από 28 εθνικά κοινοβούλια συν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μετά την ολοκλήρωση όμως και των 27 Εθνικών Κοινοβούλιο και έχω μερικά παραδείγματα εδώ με τα Δυτικά Βαλκάνια έχει υπογραφεί το 2006 και τέθηκε σε ισχύ μόλις το Δεκέμβριο του 2017. Μαρόκο το ίδιο υπεγράφει το 2006 τέθηκε σε ισχύ το Μάρτιο του 2018. Καναδάς αντίστοιχα. Και πάλι έχουμε θέμα εδώ ε, συνεχώς ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να επιταχύουν τις διαδικασίες κύρωσης γιατί πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να ολοκληρώνονται αυτά. Και πάλι το Κοινοβούλιο καμιά φορά ε, μπορεί να εκπλαγεί που του ζητούμε να δώσει τη σύμφωνη γνώμη του για συμφωνίες που έχουν υπογραφεί χρόνια πριν, γιατί περιμέναμε τα κράτη-μέλη να κάνουν τις κυρώσεις με τα κοινοβούλια πριν κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που της αναλογεί. Αυτά είναι οι συνολικές συμφωνίες. Η άλλη μεγάλη ενότητα είναι οι οριζόντιες συμφωνίες που έρχονται να ευθυγραμμίσουν και να προσαρμόσουν ε, στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο τις διμερείς συμφωνίες των κρατών μελών. Και αυτό είναι δύσκολο εγχείρημα καμιά φορά, γιατί καμιά φορά οι τρίτες χώρες αρνούνται να αναγνωρίσουν την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θέλουν να αλλάξουν τις διμερείς συμφωνίες που έχουν. Μέχρι τώρα είχαμε σχετική επιτυχία. 120 χώρες ε, το δέχτηκαν ανά τον κόσμο και έχουμε τροποποιήσει πολλές από τις διμέρειες συμφωνίες είτε με οριζόντιες συμφωνίες 50 τον αριθμό, αλλά και τα κράτη-μέλη από μόνα τους τροποποιούν τις συμφωνίες αυτές για να τις ευθεγραμμίσουν με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Πρόσφατα ολοκληρώσαμε τη συμφωνία με την Κίνα, που ήταν μια μεγάλη χώρα η οποία δεν είχε αναγνωρίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, στις συμφωνίες ως τέτοια, πολύ σημαντικό, υπογράψαμε. Ολοκληρώσαμε τις διαπραγματεύσεις πέρσι τον Οκτώβριο με την Νότια Κορέα και ελπίζουμε να υπογράψουμε πάρα πολύ σύντομα και ήδη αρχίσαμε διαπραγματεύσεις με την Ιαπωνία. Στο τέλος της διαφάνειας βλέπετε ότι εκκρεμούν ακόμα Ρωσία, Λευκορωσία, ε, Νότια Αφρική και κάποιες άλλες αφρικανικές χώρες δεν αναγνωρίζουν την δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνάπτει τις συμφωνίες. Αυτά. Μια πάρα πολύ έτσι, χονδρική ε, ε, επισκόπηση και εικόνα και να ανακεφαλαιώσω. Το 2015 παρουσιάστηκε η στρατηγική για την αεροπορία και τότε είπαμε, πήγαμε στα κράτη-μέλη και ζητήσαμε να μας δώσουν εντολή για να διαπραγματευόμαστε με άλλες χώρες. Για να επανέλθω σε μια προηγούμενη ε, διαφάνεια αυτή με το χάρτη, θα δείτε ότι τότε είχαμε ζητήσει και εντολή για να διαπραγματευτούμε την Κίνα, το Μεξικό, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία. Όταν πήγαμε στο Συμβούλιο αποφάσισαν τα κράτη-μέλη να μην μας δώσουν αυτή την εντολή. Παρόλα αυτά, μας έδωσαν εντολή για να διαπραγματευτούμε με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ε, τα οποία αρνήθηκαν να διαπραγματευτούν μαζί μας, οπότε δεν συνεχίστηκαν οι διαπραγματεύσεις και εξέπνευσε η εντολή. Έτσι έχουν τα πράγματα. Τώρα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αρχίσει ο προβληματισμός για το ποιοι είναι οι νέοι στόχοι, οι νέες χώρες για ευρωπαϊκές συμφωνίες. Στα οριζόντια θα ε, εξακολουθούμε να κάνουμε διαβήματα προς τις χώρες που δεν δέχονται την Ευρωπαϊκή Ένωση ως συνομιλητή, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε και νέες χώρες που θα ενδιαφερθούν και διάφορα στοιχεία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, κατά πόσο ενδιαφέρεται η άλλη πλευρά, τα κράτη-μέλη μας, ε, οι αγορές και πώς αυξάνεται η κίνηση των επιβατών. Όλα αυτά θα πρέπει να συνυπολογιστούν. Θα σταματήσω εδώ και με πολύ χαρά να απαντήσω σε ερωτήσεις. Merci beaucoup pour... Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσίαση που ήταν πολύ ενημερωτική, κατατοπιστική και σύντομη. Κυρία Τάλερ, ζήτησε πρώτο λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση επίσης για την γενική επισκόπηση που μας δώσατε για τα διάφορα επίπεδα συμφωνιών που υπάρχουν και που θα υπάρξουν. Έχω ένα γενικό ερώτημα ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση ο, ε, τη ανταγωνιστικότητα, της ψηφιοποίησης και της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε αυτές τις τρεις. Αυτά τα τρία επίπεδα προκλήσεων στις δικές σας διαπραγματεύσεις, πώς τις αντιμετωπίζετε, πώς τις λαμβάνετε υπόψη. Ευχαριστώ. Η κυρία Ροβέτ. Εντυπωσιάστηκα από την καταπληκτική σας ε, ε, πρόταση ότι αυτά που ε, αναφέρεται ως πλεονεκτήματα είναι όντως μειονεκτήματα αύξη πτήσεων, θέσεων. Ε, πώς όμως α, μπορείτε όλα αυτά να τα θεωρείτε πλεονεκτήματα για το πλανήτη. Πώς ζείτε σε άλλο πλανήτη. Είναι θετική αυτή η αύξηση της εναέρειας κυκλοφορίας, αυτή η αύξηση των πτήσεων με ταυτόχρονη μείωση του κόστους. Μα τα παρουσιάσετε και ως πλεονεκτήματα. Ποια θα ήταν τα ωφέλη για τον πλανήτη ο, αν μειώσουμε τις αεροπορικές μας μεταφορές. Πώς συμφωνίε αυτές θα μπορούσαν να συμβάλλουν στο μέλλον, όπου στόχος μας δεν θα είναι η αύξηση των αεροπορικών μεταφορών, αλλά η μείωση της ενέργεια κυκλοφορίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ροβέτο. Ο κύριο Κόφ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Να, όντως, ε, κάναμε μια παραλλαγή της προηγούμενη ερώτηση Στον αιώνα είχαμε αυτό το όραμα της απεριόριστης επέκτασης, αλλά τώρα προσκρούμε στην περιβαλλοντική πραγματικότητα και τους περιορισμούς ε, του πλανήτη ως προς την επέκτασή του. Και τι γίνεται με τις συμφωνίες αυτές. Υπάρχει κάποιο περιθώριο για περιβαλλοντική δράση στα πλαίσια των ε, συμφωνιών αυτών. Τι γίνεται με τα καθόλου ζητήματα των δρομολογίων, των εξοικονόμησης, ε, καυσαερίων, τη, τα δρομολόγια που παίρνουν από διάφορες χώρες. Επίσης, τι κόστος ε, και τι τέλη ε, περιμένετε από τα κράτη-μέλη και πώς τα κατανέμετε. Πάντως, ο λέφτος στο δωμάτιο είναι αυτό που είδαμε την περασμένη Παρασκευή στους δρόμους, στα συλλαλητήρια. Σίγουρα σας δεσμεύει η ισχύουσα νομοθεσία και σας περιορίζει. Αλλά υπάρχει κάποια δυνατότητα, κάποιο περιθώριο να λάβετε υπόψη τις συμφωνίες αυτές και τη μεγάλη πρόκληση να μειώσουμε το διοξείδιο του άνθρακα. Φαίνεται δεν έχουμε και μεγάλη πιστοσύνη στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είπε ότι η αεροπορία θα θα ενταχθεί στο σύστημα εμπορίας εκπομπών. Μακάρι, το ευχόμαστε. Αμήν και πότε. Μην γελάτε, γιατί τώρα χαμογελάτε, αλλά ήταν μια επίσημη αναγγελία τη υποψήφια πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπει αεροπορία στο σύστημα εμπορία εκπομπών. Δεν ξέρω πώ θα τα καταφέρει, αλλά εσεί ε, και η γενική σα διεύθυνση έχετε γνώμη για το θέμα αυτό. Άλλε ερωτήσει, Ρικέ, Λεσαντό, Γκαρσία, όχι. Ναι ή Όχι, οπότε παρακαλώ τον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Ο γενικός στόχος ε, για τις εκπομπές είναι κοινός για όλους μας δεν σημαίνει απαραίτητα μείωση των αεροπορικών ταξιδιών. Στόχος πρέπει να είναι μείωση των εκπομπών που, προκαλεί, που προκαλούν τα αεροπορικά ταξίδια. Εκεί βρισκόμαστε και συμφωνούμε. Δεν υπάρχει διχογνωμία εδώ μεταξύ των όσων είπε νέα πρόεδρος και των ε, πραγμάτων που θα υλοποιηθούν κατά την εντολή της, κατά τη θητεία της, το τι κάνουμε εμείς ε, σε διεθνές επίπεδο γενικότερα. Παρεπιπτόντως, οι συναδελφοί μας σήμερα βρίσκονται στο Μόντρεαλ, στην ΚΑΟ, για να μελετήσουν στην ΚΑΟ, για να συζητήσουν ακριβώς αυτό το μείωση των εκπομπών. Οπότε ο στόχος είναι κοινό, είναι ο ίδιος. Τι μπορούμε να κάνουμε στις συμφωνίες αεροπορίας, ανεξάρτητα από το τι θα κάνουμε στην ΚΑΟ, και με τα αναλλακτικά καύσιμα, με τα πιο αποδοτικά αεροπλάνα ή με καλύτερο σχεδιασμό των διαδρομών τι κάνουμε σε αυτές τις συμφωνίες. Δεν μιλάμε μόνο για δικαιώματα κυκλοφορίας. Ε, μελετάμε μια πλατφόρμα συνεργασίας. Έχουμε ένα άρθρο σε αυτές τις συμφωνίες για το περιβάλλον με στόχο τη συνεργασία για θέματα κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα του περιβάλλοντος και έχουμε και μηχανισμό για αυτό. Επίσης έχουμε τη δυνατότητα καλύτερης συνεργασίας για να έχουμε πιο απευθείας ευθείες ε, διαδρομές. Ξέρετε εσείς με το ETM ε και το SESO υπάρχει δυνατότητα να υπάρχουν όσο το δυνατόν πιο ευθείε πτήσει ε, και σύντομε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό γίνεται και σε διεθνέ επίπεδο. Αυτό γίνεται με τη συνεργασία με αυτέ τι χώρε σε διάφορου τομεί. Οι συμφωνίε αυτέ λοιπόν δεν είναι αυτέ καθεαυτέ η απάντηση στα ζητήματα, αλλά ένα στοιχείο που συμβάλλει στο να επιτευχθούν αυτοί οι κοινοί στόχοι. Ωραία. Εγώ έχω μια ερώτηση επειδή θα έχουμε τη Γενική Συνέλευση του ΙΚΑΟ. Σήμερα η Ευρώπη δεν θεωρείται ότι θα πρέπει να ηγηθεί του ζητήματος των εκπομπών και να δείξει μεγαλύτερη φιλοδοξία από τον ΙΚΑΟ, ο οποίος ΙΚΑΟ δεν φαίνεται να προχωρά. Η Ευρώπη χρειάζεται μεγαλύτερη φιλοδοξία. Οπότε να μην αφήνει την αποκλειστικότητα των εκπομπών στον ΙΚΑΟ. Ίσως να μην έχετε το δικαίωμα να μιλήσετε γι' αυτό, αλλά ταυτόχρονα εγώ πιστεύω ότι η Ευρώπη είναι βρίσκεται στην κατάλληλη χρονική στιγμή, την οποία πρέπει να αξιοποιήσει. Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ηγείται, πιστεύω, στο Μόντρεαλ, στο Νικάο. Και όλοι συμφωνούμε ότι τα προβλήματα της αεροπορίας είναι παγκόσμια. Δεν μπορούν να επιληθούν σε μια γωνιά του κόσμου. Χρειαζόμαστε μια παγκόσμια λύση. Ταυτόχρονα έχουμε συνείδηση του ότι η λύση αυτή θα πρέπει να είναι ανθεκτική, αποδοτική αυτό κάνουμε αυτέ τι μέρε στον ΙΚΑΟ. Θα δούμε τι θα γίνει σε εκείνο το επίπεδο του ΙΚΑΟ και μετά θα αποφασίσουμε τι θέλουμε ή όχι σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν άλλε ερωτήσει. Όχι. Ευχαριστούμε πολύ, αξιότιμε κύριε, που μας εφήρωσε το χρόνο σας. Ελπίζω να μας έρχεστε πιο συχνά. Υπό τα διάφορα δεν έχουμε τίποτα. Η επόμενη μας συνεδρίαση θα λάβει χώρα στις 6 Νοεμβρίου. Στις 9 το πρωί ακριβώς. Και θα συνεχιστεί και το απόγευμα τέλος της συνεδρίασης, αλλά δεν έχει τελειώσει η μέρα μας γιατί έχουμε τη συνεδρίαση των συντονιστών στις 5. Διάλειμμα λοιπόν 20 λεπτών. Ευχαριστώ.